Good morning, everybody. Καλημέρα σε όλους. Θα αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Καλημέρα και στα Ισπανικά, λέει η Πρόεδρος. Θα αρχίσουμε με την σημερινή μας συνεδρίαση. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη που είναι το πρώτο σημείο. Δεν ξέρω αν έχει κάποιος κάτι να πει για την ημερήσια διάταξη, αλλιώς θεωρείται εγκεκριμένη. Σύμφωνοι. Ωραία. Εγκρίνεται και συνεχίζουμε. Έγκριση των πρακτικών. Τα πρακτικά τα έχετε, είναι στη διάθεσή σας. Αν έχετε κάποια παρατήρηση, Παρακαλώ να μου την πείτε. Όχι. Σημείο 3. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Στις ανακοινώσεις της Προέδρου πρέπει να σας πω ότι το χρονοδιάγραμμα για την έκθεση όσον αφορά τις οικιακές βοηθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει έχετε στα χαρτιά σας το νέο χρονοδιάγραμμα. 15 Οκτωβρίου θα εξεταστεί η έκθεση και 13 Νοεμβρίου θα έχουμε τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στις 14 Ιανουαρίου στην Επιτροπή μας και στη δεύτερη σύνοδο του Φεβρουαρίου θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Όσον αφορά τώρα την αποστολή μας στην Ιρλανδία, 24 και 25 Σεπτεμβρίου. Οι συντονιστές έχουν αποφασίσει σχετικά, το έχουμε συζητήσει με όλες τις πολιτικές ομάδες και τελικά αποφασίσαμε 10 μέλη να συμμετέχουν, 8 βάση ποσοστώσεων, συν την πρόεδρο και κάποιον από την Ιρλανδία την ίδια. Αυτές είναι οι ανακοινώσεις της Προέδρου που είχα. Συνεχίζουμε λοιπόν και περνάμε τώρα στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Θα συζητήσουμε για την έκθεση τη σχετική με τις γυναίκες στον επιστημονικό και πανεπιστημιακό χώρο και η όρατη φραγμή που αυτές αντιμετωπίζουν. Αυτό είναι το θέμα. Η συγγήτρια, η κυρία Βόζαμπερκ, έχει το λόγο λοιπόν και μετά θα συζητήσουμε με παρεμβάσεις από τους σκιώδεις εισηγητές και τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Παρακαλώ κυρία Βόσμπερ και σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πω ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια όταν ασχολούμαι με ένα αντικείμενο όπως αυτό που ε, υπάρχει στην έκθεση που μου έχει εμπιστευτεί η Επιτροπή. Να πω γιατί η διότι από τα 30 χρόνια της μάχημης δικηγορίας έχω ασχοληθεί ειδικά με δικαιώματα γυναικών στον επαγγελματικό τομέα και εννοώ σε επίπεδο γυναικών καριέρας, γυναικών που βάζουν στόχους και έχουν την δυνατότητα και την ικανότητα, αλλά σε μεγάλο βαθμό, σε όλα τα κράτη-μέλη παρατηρείται το φαινόμενο, εμποδίζονται να πετύχουν αυτούς τους στόχους λόγω των εγγενών αδυναμιών που υπάρχουν στις αντιλήψεις, στα στερεότυπα και σε παγιωμένες νοοτροπίες, οι οποίες κάθε άλλο παρά τιμούν την δημοκρατία και τις, ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα για τα οποία παλεύουμε μια ολόκληρη ζωή. Στην έκθεση, όπως θα έχετε δει, προσπαθούμε να επικεντρωθούμε σε ένα αντικείμενο και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει σε μεγάλο βαθμό. Αυτό θα φανεί κατά πόσον ομόφωνα ή σε μεγάλη πλειοψηφία ψηφιστεί αυτή η έκθεση. Ακριβώς να εστιάσουμε γιατί έχουμε φτάσει στο 2015 και ακόμη μιλάμε για εμπόδια, στη, τη γυάλινη οροφή όπως λέγεται, το glass ceiling, για εμπόδια στην εξέλιξη των γυναικών στις επιχειρήσεις, στο πανεπιστήμιο, στην ακαδημαϊκή δηλαδή καριέρα, στα κέντρα έρευνας, σε εκεί όπου πραγματικά το γυναικείο μυαλό έχει αποδείξει, επί ίσης με το ανδρικό, ότι είναι εξαιρετικά δημιουργικό και παραγωγικό. Αυτά τα εμπόδια προσπαθεί αυτή η έκθεση να τα αντιμετωπίσει επιχειρώντας και με το σύνολο των τροπολογιών να μην μείνει σε ένα θεωρητικό επίπεδο αλλά να προτείνει ένα βήμα παραπάνω γιατί ο στόχος δεν είναι απλώς να παρεμποδίσουμε την εξέλιξή τους ή σε κάποιο βαθμό να μειώσουμε αυτά τα εμπόδια αλλά ή δυνατόν να τα εξαλείψουμε Φυσικά δεν φιλοδοξώ η έκθεσή μας να, αυτομάτως να μπορεί να εξελίψει. Αυτό πρακτικά δεν γίνεται. Αλλά σίγουρα με θετικές κατευθύνσεις σε ένα στόχο που βάζουμε και τον υπηρετούμε όλοι, ανεξάρτητα από ποια πολιτική ομάδα προερχόμαστε, ποιες αντιλήψεις υπηρετούμε, νομίζω ότι ακριβώς ο στόχος αυτής της έκθεσης είναι κοινό. Γιατί αλλιώς δεν θα βρισκόμασταν εδώ, δεν θα υπηρετούσαμε τέτοιες αξίες μέσα σε αυτή την Επιτροπή να σας ενημερώσω ότι ε, έχουμε 114 τροπολογίες, εκ των οποίων σε 10 έχουμε συμβιβαστική κατεύθυνση. Είναι 10 οι συμβιβαστικές τροπολογίες όπως τα είδατε και είναι συμβιβαστικές διότι παρά το γεγονός ότι προέρχονται όλες οι προστιθέμενες αξίας ε, αντιλήψεις έχουν κατατεθεί από διαφορετικές αφετηρίες, σκέψεις, τίνουν στον ειδικό σκοπό που υπηρετεί αυτή η έκθεση. Και εννοώ, παραδείγματο χάρη, γιατί να υπάρχουν γυναίκες που υπηρετούν ε, υψηλά αξιώματα και δεν αμείβονται επίσης όρεις με αντίστοιχους άντρες όταν έχουν αντικειμενικά, ουσιαστικά και τυπικά προσόντα τα ίδια. Γιατί αυτό στα κράτη-μέλη δεν έχει ρυθμιστεί με τις εθνικές νομοθεσίες. Γιατί εκεί υπάρχει όπως ξέρετε η αρχή της επικουρικότητας. Αλλά και εμείς βάζουμε το λιθαράκι να κατευθύνουμε τις εθνικές νομοθεσίες έτσι ώστε επίσης ώρες να αντιμετωπίζονται αυτά τα κορυφαία θέματα. Επίσης, γιατί ε, να μην έχουμε κατορθώσει τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, βάζω παραδείγματα, να μπορέσουν να προάγουν και να προωθούν ιδιαίτερα στη νεολαία όπου, και ιδιαίτερα στον τομέα της εφηβείας όπου αναπτύσσονται οι προσωπικότητες εκείνα τα πρότυπα και στερεότυπα που πραγματικά οδηγούν τις νέες γυναίκες που έχουν θέληση και ικανότητες να μπορέσουν να κατακτήσουν αυτό το οποίο επιδιώκουν. Ε, επιπρόσθετα να σας πω ότι οι αρνητικές ψήφοι τις οποίες θα δείτε ότι προτείνουμε δεν ε, ε, ας πούμε στρέφονται επικριτικά σε αυτές τις τροπολογίες γιατί έχουν προστιθέμενη αξία, έχουν πολύ σημαντικά έχουν συμβάλει στην έκθεση. Είναι αρνητικές διότι ουσιαστικά φεύγουν από το σκοπό που υπηρετεί η έκθεση. Το να, παραδείγματος χάρη, το να προτείνουμε μια τροπολογία η οποία ε, ενισχύει την ανάγκη της κατοχύρωσης της ισότητας, εκφεύγει από το εξειδικευμένο αντικείμενο της ισότητας σε συγκεκριμένους τομείς, σε ειδικέ ε, βαθμίδες επιστήμης, σε ειδικά πόστα της εξέλιξης, στην επιχειρηματικότητα και στην κατάκτηση εκείνων των τομέων ευθύνης για τους οποίους ορθώνονται τα εμπόδια. Αυτό είναι που πολεμούμε. Ε, στο τέλος να, να σας ενημερώσω ότι υπάρχουν και τρεις ε, προφορικές ε, τροπολογίες που προέρχονται από τον σκιώδη συνεισηγητή μας θα έλεγα εγώ, όχι σκιώδη εισηγητή, οι εισηγητές από κοινού εργάζονται, τον κύριο Σεμπαστιά που με χαρά τις φιλοξενούμε αυτές. Τέλος, σε αυτή την σύντομη έτσι αναφορά μου θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς την advisor την Ντανιέλα Σένκα από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τη Ζουζάνα ε, Χρούσκοβα, πάντα μπερδεύομαι στο όνομα Ζουζάνα μου, από τη Γραμματεία της Επιτροπής ΦΑΜ, διότι η παρουσία του στη σύνταξη πραγματικά της έκθεσης είναι, δεν είναι συμβολική, είναι εξαιρετικά σημαντική αυτό το οποίο διακρίνει πάντοτε τις εργασίες της Επιτροπής μας είναι η συλλογικότητα και μπορεί την πρώτη ευθύνη να έχει ένας εισηγητής, αλλά αν δεν συμπράττουν σε θετική κατεύθυνση και οι συνεισηγητέ, δηλαδή οι σκιώδεις εισηγητές και βεβαίως η τεχνική εξειδικευμένη υποστήριξη, ποτέ μια έκθεση δεν έχει αρτιότητα. Με αυτές τις λίγες σκέψεις θα ήθελα να παρακολουθήσω τη συνέχεια της συζήτησής μας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Βόζεμπερτ. Τώρα θα δώσω το λόγο στους κοιόδης συζητητές των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Ποιος θα αρχίσει. Παρακαλώ κύριο Σεμπάστιαν. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ την εισηγήτρια για τα καλά της λόγια και κυρίως για την προσπάθεια που κάνει προκειμένου η έκθεση αυτή να προχωρήσει. Είναι πολύ σημαντική και υπάρχει μεγάλη ευρεία συνένεση από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα στην πρώτη συζήτηση που κάναμε για αυτό το θέμα. Εμείς προσπαθούμε να ζητήσουμε και εμείς αυτή την αλλαγή, όπως ζητάει και η συγκήτρια, αυτή την αλλαγή νοοτροπίας όσον αφορά τις ευθύνες στην οικογενειακή ζωή. Διότι η γυναίκα που επαγγελματικά βρίσκεται στην έρευνα αντιμετωπίζει αυτούς τους αόρατους φραγμούς γιατί θεωρείται ότι στην οικογενειακή ζωή, η μέρημνα των παιδιών, όλα αυτά είναι δικιά της δουλειά. Είναι ένα κλισέ αυτό που πρέπει να αλλάξει. Και γι' αυτό λοιπόν θελήσαμε με τις τροπολογίες μας να τονίσουμε αυτό ακριβώς το στοιχείο. Ευχαριστώ πολύ επίσης την εισηγήτρια που δέχτηκε τις δικές μας τροπολογίες που έφτασαν και λίγο αργά. Ξέρω ότι εγώ φταίω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, δεν έχω καμία δικαιολογία. Εγώ έκανα λάθος στην ημερομηνία στις προθεσμίες, οπότε ζητώ συγγνώμη, δεν θα ξανασυμβεί. Αυτά να πω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από το γενικό αποτέλεσμα και ελπίζω να υπάρχει ομοφωνία, η σημαντική πλειοψηφία. Πιστεύω ότι μπορούμε να στηρίξουμε αυτό το έργο και από εδώ και πέρα να δουλέψουμε όλοι σοβαρά, ώστε στα σοβαρά να πάρουν όλα τα θεσμικά όργανα τα όσα περιλαμβάνει η έκθεση αυτή. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Σεμπαστιά. Η κυρία Αντσίλα έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφό μας κυρία Βόζενμπεκ και για το κείμενο της εκθέσεως και για την πολύ θετική συνεργασία. Είναι καλή η παρουσίαση του θέματος, καλή η αντιπαράθεση ας πούμε με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον επιστημονικό και πανεπιστημιακό τομέα. Στην εξέταση των τροπολογιών διατυπώνουμε ότι θα θέλαμε προτείνουμε δηλαδή, καλύτερη διασύνδεση μεταξύ πανεπιστημιακού τομέα και μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Καθώς και στο τοπικό επίπεδο για τις γυναίκες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε επιστημονικούς τομείς, αυτή η κίνηση να βελτιωθεί. Έχω καταθέσει τροπολογίες, ευχαριστώ που τις δέχθηκε η, η και αναφέρομαι ιδίω σε θέσπιση βραβείων για γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον επιστημονικό τομέα. Αυτά τα βραβεία μπορούν να δίνονται από επιχειρήσεις ή από άλλους φορείς για επιτυχίες στον επιστημονικό τομέα που πιστώνονται σε γυναίκες. Η συνάδελφός μου εξάλλου, εξάλλου είπε όλα όσα χρειάζεται για την εξήγηση και ευχαριστώ και εγώ για τις τροπολογίες των συναδέλφων. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μιλάντα, έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγητρία και πάλι για τη δουλειά της, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το ζήτημα που συζητούμε, γυναίκε και επιστήμη, δεν είναι απλό. Ήδη αναφέρθηκε. Είναι περίπλοκο λόγω χάρη ο αρνητικό αντεκτυπό των στερεοτύπων σε σχέση με τα φύλλα, είναι κάτι που το αντιμετωπίζουμε διαρκώ και σε αυτό το πλαίσιο και έντονα. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω μια πτυχή αυτή τη έκθεση. Ω επικοδομητική συνεισφορά. Πιστεύω ότι ο κατάλογο ψηφοφοριών που έχουμε μπροστά μα περιλαμβάνει συμβαστικέ τροπολογίε και τροπολογίε που δεν σχετίζονται αυστηρώ με το κάθε αυτό θέμα τη έκθεση. Πιστεύω λοιπόν ότι αν θέλουμε να είμαστε συνεπεί στη δουλειά μα ω Επιτροπή ΦΑΜ που είναι ήδη αρκετά περιπλοκή, θα πρέπει να φροντίσουμε και να είμαστε πολύ ακριβεί και στοχευμένοι στο αποτέλεσμα του ψηφίσματο για την Ολομέλεια. Ευχαριστώ. Muchas gracias. Ευχαριστούμε. Τέλος. Η κυρία Γκέρλινγκ έχει το λόγο για αυτόν τον γύρο παρεμβάσεων. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Όταν ε, αρχίσαμε να δουλεύουμε πάνω στην έκθεση αυτή για τους όρατους φραγμούς, την γυάλινη οροφή όπως την ονομάζουμε, πιστεύοντας ότι είναι το τελευταίο, ο τελευταίος φραγμός, τον οποίο δεν μπορεί να ξεπεράσει κανείς, διαπιστώσαμε ότι και προηγουμένως υπάρχουν άλλα διάφορα στρώματα με τέτοια ώρα τα εμπόδια πριν φτάσουμε σε αυτό το τελευταίο. Στην επιστήμη, γυναίκες μηχανικοί, χρειάζονται βοήθεια. Το ζήτημα λοιπόν είναι τι θα έπρεπε να γίνει, τι, πώς θα έπρεπε να διαμορφωθεί μια τέτοια βοήθεια Σίγουρα χρειάζεται αλλαγή στην οτροπία, στις προσδοκίες, αλλά χρειάζεται και αλλαγή στην ομοθεσία. Πολλές φορές πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες να ακολουθήσουν και να κάνουν αυτό που θέλουν. Ήμουν σε ένα γάμο πριν από μερικές εβδομάδες. 28 ετών, PhD είχαν εκεί δύο που παντρεύτηκαν και οι δύο μηχανικοί, έξυπνοι άνθρωποι, έξυπνα παιδιά, αεροναυπηγικοί. Και τους κοίταζα και σκεφτόμουν σε 10 χρόνια πού θα βρίσκονται σε 15 χρόνια αυτοί, ποιος από τους δύο θα τα καταφέρει καλύτερα στην καριέρα του, ποιος, ε, ποιον η δουλειά θα αξιολογηθεί περισσότερο. Η νύφη είπα μάλλον στην ύφη, ενημέρωσε με, θα ήθελα πολύ να ξέρω πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα, πώς θα πάνε οι καριέρες σας. Οι γυναίκες δηλαδή υπάρχουν με προσόντα, με πολύ δυνατά προσόντα και με προθέσεις να προχωρήσουν, αλλά κάτι παστραβά τελικά στη διαδρομή. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση με τις εκθέσεις αυτές πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται και στις χώρες μέλη και εγώ αισθάνομαι άσχημα διότι μόνο 7% στον τομέα ακριβώ αυτού του κλάδου είναι γυναίκες. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι οι γυναίκες θα έχουν καταφέρει καλά στο Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον μόνο 7% σε αυτό τον κλάδο είναι γυναίκες, είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει η κυβέρνησή μου, πρέπει να το κοιτάξει και να κάνει κάτι. Συνεπώς, πού βρισκόμαστε. Θέλω εθάρρυνση για τις γυναίκες που μπαίνουν σε κλάδους που παραδοσιακά θεωρούνται αδρικοί. Πρέπει να τις ενθαρρύνουμε. Έχουν την πρόθεση οι γυναίκες και η ομάδα μου χαίρομαι πολύ που μπορεί να στηρίξει αυτή την έκθεση. Κάπου έχουμε κάποιες δυσκολίες. Για παράδειγμα, δεν είμαι σίγουρη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης έχει να προσφέρει πολλά. Και συμφωνώ νομίζω με τους συναδέρφους από την Άλντε πρέπει να επικεντρωθούμε σε την πειθαρχία και να έχουμε κοινέ κατευθυντήριε γραμμέ για τα πανεπιστήμια. Και αυτό δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναμειχθεί σε αυτό. Δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει. Τι χώρε μέλη πρέπει να ενθαρρύνουμε να το κάνουν. Και δεν θέλω ένα ευρωπαϊκό ταμείο ε, συνταξιοδοτικό εδώ. Δεν βλέπω τι δουλειά έχει. Κατά τα άλλα, ευχαρίστω η ομάδα μου θα στηρίξει την έκθεση αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τέλος, η κυρία Κοσλόφσκα. Αυτή είναι η τελευταία σε αυτό το γύρο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, επιθυμώ και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε το θέμα. Βεβαίω είναι λυπηρό διότι στον 21ο αιώνα εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η κρυστάλλινη οροφή. Σε όλους τους τομείς, στην επιστήμη, στις business, στον αθλητισμό, ακόμα και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς υπάρχει η κρυστάλλινη οροφή. Προετών στην Πολωνία είχα ασχοληθεί με το θέμα αυτό, ιδίω ε, στον χώρο των επιστημών και εξέτασα τι γίνεται στην Πολωνική Πανεπιστημιακή Επιτροπή, έτσι ονομάζεται ο θεσμός αυτός, και διεπίστωσα ότι αυτό το όργανο υψηλωτά του επίπεδου με ανθρώπους με εξαιρετικά προσόντα απαρτίζεται σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες. Μέσα σε 100 ονόματα μόνο 4 γυναίκες. Και εγώ ήμουν επιστημονική συνεργάτης και εγώ έχω διδακτορικό και γνωρίζω ότι στα διδακτορικά ακόμα το ποσοστό είναι 50%-50%. Στο επίπεδο πλέον των καθηγητών και καθηγητριών το, επίπεδο, το, ε, ποσοστό των γυναικών φτάνει τα 20%. Και όμως, όπως σας είπα, στο υψηλό αυτό επίπεδο της ε, Επιτροπής Επιστημών το ποσοστό των γυναικών ήταν 4%. Και διερωτήθηκα σε τι οφείλεται αυτό. Σας τα λέω αυτά κάπως ανεκδοτολογικά, γιατί αυτή η κατάσταση ανεβρίσκεται παντού και δεν είναι μόνο θέμα νομικών διατάξεων. Και στην Πολωνία έχουμε ψηφίσει κώδικα διοντολογίας που λέει ότι δεν επιτρέπονται διακρίσεις, πρέπει πάντοτε να προκυρήσουν οι θέσεις είτε για άνδρες είτε για γυναίκες, δηλαδή να απευθύνονται και στα δύο φύλλα, αλλά αυτά από μόνα τους δεν αλλάζουν την νοοτροπία, την πολιτιστική ας πούμε στάση, ή αλλάζει για λίγο και μετά επανέρχονται. Θυμηθείτε και την Τινησία και άλλες χώρες, όπου κάτι σκυρτά, κάτι κινείται, η διάρκεια όμως είναι πολύ σύντομη. Και όσες πρόοδοι επιτυγχάνονται, επιτελούνται, μετά δυστυχώς χάνονται ξανά. Ανεξαρτήτως λοιπόν τώρα των διατάξεων του εργατικού δικαίου, εκεί που πρέπει να στοχεύσουμε είναι η αλλαγή των νοοτροπιών. Εγώ είχα δραστηριοποιηθεί και στο Πολωνικό Κοινοβούλιο και εκεί ασχολήθηκα με μελέτη επιστημονικών θεμάτων και είδα ότι στα επιστημονικά όργανα, στους επιστημονικούς φορείς δεν υπάρχουν καθόλου γυναίκε. Κάποτε είχαμε σκεφτεί και εμεί να βάλουμε ποσοστώσει. Είπαμε δεν είναι δυνατόν να επιλέγονται μόνο άνδρε. Αντιμετωπίσαμε ωστόσο μια λυσαλέα αντίδραση που οδήγησε τελικά στο να μην εγκριθεί η νομοθεσία αυτή. Όταν λοιπόν συζητούμε τέτοια θέματα, γρήγορα αποδείχνεται ότι δεν υπάρχει πραγματική ισότητα, διότι υπάρχει μια πεποίθηση η οποία αποκλεί τις γυναίκες. Και μόνο μέσα από την οδό του δικαίου δεν αντιμετωπίζει το θέμα. Χρειάζεται να αλλάξουν τα μυαλά, χρειάζεται να αλλάξουν οι νοοτροπίες. Κάθε συζήτηση, κάθε άκραση απόψεων που συντελεί προς αυτή την κατεύθυνση είναι καλοδεχτή. Ευχαριστούμε. Η συγκίτρια τώρα. Θέλει κάτι να πει για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ε, απλώς να προσθέσω, κυρία Πρόεδρε, καταρχάς ευχαριστώ τους σκιώδεις εισηγητές για τις τοποθετήσεις του σε πρώτο επίπεδο. Ήθελα να, κλείνοντας να προσθέσω, συμφωνώ απόλυτα, νομίζω όλες συμφωνούμε, όλες και όλοι συμφωνούμε, σε αυτό το οποίο στην τελευταία απόχρωση της φωνής της κυρίας ε, ε καλά το είπα, <laughs> ότι το πρόβλημα υπάρχει διότι παρά το γεγονός ότι στα κράτη-μέλη οι νοοτροπίες είναι διαφορετικές των λαών μας, έχουν διαφορετικές ιστορικές καταβολές, διαφορετικό ταπεραμέντο, διαφορετικό τρόπο σκέψης. Ειδικά σε αυτό το νοσηρό φαινόμενο συμπίπτουν. Υπάρχουν δηλαδή σε όλα τα κράτη-μέλη νοσηρές νοοτροπίε, οι οποίε παγιώνονται και συνεχίζονται και εμποδίζουν, δηλαδή μάλλον ενισχύουν αυτό το φαινόμενο το οποίο η έκθεση προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Οι νοοτροπίε όμως, για να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, αντιμετωπίζονται ριζικά με δράσεις κάτω από δύο φυτόρια. Το ένα είναι η οικογένεια και το άλλο είναι η παιδεία και μάλιστα η μέση εκπαίδευση. Αν λοιπόν καλλιεργούνται οι νοοτροπίες με, αυτά, με αυτές τις δύο κατευθύνσεις αρχίζουν και ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης, διότι να πούμε ότι πέραν από τα εμπόδια τα οποία εμείς πολεμούμε σε αυτή την έκθεση, υπάρχει και μια ανατροπή ως προς τους στόχους που βάζουν πολλές γυναίκες, γιατί πιστεύουν απριόρι ότι δεν πρόκειται να τους πετύχουν επειδή υπάρχουν αυτές οι νοοτροπίες. Και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Με δράσεις λοιπόν συγκεκριμένες, βήμα-βήμα, οι νοοτροπίες δεν αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλάζουν όμως αν υπάρχει μια συστηματική οδός και συμφωνώ ότι δεν μπορεί μόνο με μια νομοθεσία από κάθε κράτος μέλος να αλλάξει νοοτροπία. Θέλει ε, διαδραστικότητα, πολλές δράσεις σε πολλά επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση με την έκθεση αυτή φιλοδοξούμε να βάλουμε ένα ε, ουσιαστικό λιθαράκι στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βόζεμπεργκ. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σήμερα όταν ολοκληρώσουμε τις συζητήσεις και την ψηφοφορία για τα άλλα θέματα. Και περάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η γνωμοδότηση για το Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Οικονομικό έτος 2016. Η συντάκτρια κυρία Ματέρα δεν ε, μπορούσε να είναι εδώ σήμερα, οπότε η κυρία Πετή θα πάρει το λόγο στη θέση της. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα αναλάβω να παρουσιάσω την έκθεση εκ μέρου τη κυρία Ματέρα, η οποία ε, ζητά συγγνώμη που δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας. Είναι η υπεύθυνη εισηγήτρια για το δημοσιονομικό έτος 2016. Πρόκειται για μία έκθεση η οποία απευθύνεται στην Επιτροπή Προπολογισμών. Η κυρία Ματέρα ε, θεώρησε πολύ σημαντικό να εργαστεί επί του θέματος αυτού, διότι έτσι όλες οι προτεραιότητες μας ως προς τον προπολογισμό μπορούν να ενσωματωθούν στο τελικό σχέδιο. Δεδομένου ότι υπάρχουν ανισότητες μεταξύ των διαφόρων κατων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Ματέρα θεωρεί ότι είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι οι ίσες ευκαιρίες θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάλυση της αρχής ισότητας των φύλων και του πώς αυτή αντικατοπτρίζεται στον προπολογισμό θα πρέπει να διέπει κάθε σημείο του προπολογισμού. Τέσσερα είναι τα βασικά σημεία. Πρώτα απ' όλα η ανάγκη να προβλέψουμε πόρους για να ενισχύσουμε τη θέση των γυναικών στις επιστήμες, την παιδεία και την αγορά εργασίας, έπειτα να ε, διευκολύνουμε τις ε, επιχειρηματικές πρωτοβουλίες των γυναικών, να ε, διατηρήσουμε το πρόγραμμα Δάφνη και επίσης να προβλεφθούν χρηματοδοτικά μέσα για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ισότητα των Φύλων και το ίδιο για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για να παρακολουθούνται οι μορφές βίας κατά των γυναικών. Η κυρία Ματέρα ευχαριστεί όλους τους ε, συναδέλφους για τη συνεργασία τους και αν έχετε ερωτήσεις μπορείτε να απευθείτε στους συνεργάτες της, στους βοηθούς της ή στην ίδια προσωπικά. Θα απαντήσει μέσω μηνύματος. Ευχαριστούμε πολύ. σκιώδε τώρα. Ποιος θέλει το λόγο? κύριος Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους της Μόνικα Βάνε που είναι υπεύθυνη από την ομάδα μας για την έκθεση αυτή και που δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ. Εκ μέρους της θέλω να μιλήσω. Εμείς υποβάλλουμε μια τροπολογία γιατί η πρόταση του Συμβουλίου να μειώσει τα χρήματα που πάνε στην ε, προώθηση της ισότητας και της μη διάκρισης έχουν μειωθεί. Λοιπόν, ξέρουμε ότι είμαστε σε κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γι' αυτό ακριβώ είναι πολύ σημαντικό να στοιχηματίζουμε ακόμα περισσότερο σε τέτοιου είδους πολιτικές, γιατί οι γυναίκες είναι τα κύρια θύματα, όπως γνωρίζουμε, της κρίσης. Συνεπώς, η συνάδελφος έχει δουλέψει πάνω σε αυτήν την τροπολογία με την οποία ζητάει να ληφθεί υπόψη το θέμα των δύο φύλων στον προπολογισμό συστηματικά με συγκεκριμένες παραμέτρους γιατί είναι βασικό στοιχείο, βασικό εργαλείο όχι μόνο υπέρ της ισότητας των δύο φύλων, αλλά και για να καταπολεμήσουμε την κρίση αυτή η οποία πλήττει όλος ιδιαίτερο τις γυναίκες στην Ευρώπη. Αυτά έχουμε να πούμε και ελπίζουμε να περάσει η άποψή μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Σεμπαστιά. Συνεχίζουμε Περνάμε στο επόμενο θέμα. Είναι η γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ο κύριος Ελτασούν, τώρα φτάνει, οπότε μας ζήτησαν αν μπορούμε να αλλάξουμε τη σειρά των εκθέσεων προς συζήτηση. Η κυρία Χόνιμπολ, από ό,τι βλέπω, είναι εδώ. Οπότε μπορούμε να συζητήσουμε πρώτα την ε, γνωμοδότηση στην Επιτροπή Λίμπε όσον αφορά την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά τη μετανάστευση. Κύριε Χόνιμπολ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ευκαιρία να σας παρουσιάσω την γνωμοδότησή ε, μου. Έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων σήμερα δεν υπάρχει τίποτε που να έχει συνταχθεί ακόμη πέραν από την ίδια την γνωμοδότηση. Οπότε, ό,τι έχω γράψει είναι οι δικέ μου ιδέε, χωρί να ξέρω ακριβώ πώ θα το τοποθετηθούν άλλε επιτροπέ όπω η Λίμπερ. Τα βασικά σημεία τώρα. Η κατάσταση των γυναικών και κοριτσιών στην Μεσόγειο, ιδίω μεταξύ των ετούντων άσυλο, Ξέρουμε πόσο απέσια είναι όσα συμβαίνουν, δεν θέλω να περάσω σε λεπτομέρειες, απλώς αυτό, αυτό που βλέπουμε Αυτό που βλέπουμε είναι ένα τεράστιο, το, το μεγαλύτερο κύμα μεταναστών προς την Ευρώπη από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό δείχνει το μέγεθος και τις διαστάσεις αυτής της κρίσης. Είναι λοιπόν σαφές το τι συμβαίνει και χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη στρατηγική απόκριση σε αυτό το φαινόμενο. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει μακροπρόθεσμα και πώς το φαινόμενο αυτό θα εκδηληφθεί και στο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιτόπου ώστε να βεβαιωθούμε ότι η θέση των γυναικών και κοριτσιών λαμβάνεται υπόψη. Προς στιγμήν αυτό δεν συμβαίνει. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία για το θέμα της ισότητας των φύλων στον τρόπο που τα μεταχειριζόμαστε τα ε, ζητήματα αυτά. Στην Επιτροπή λοιπόν γυναικών πρέπει να δούμε ακριβώ τι συμβαίνει με τι γυναίκε και τα κορίτσια, διότι ενδεχομένω αυτέ να υποφέρουν περισσότερο από του υπόλοιπου πρόσφυγε. Είναι πιο ευάλωτε σε αυτέ τι συνθήκε. Και το ίδιο και για την συνέχεια τη πορεία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το πώς τα κάτι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση μεταχειρίζονται το τους σε άσυλο και πώς βλέπουν το ζήτημα του ασύλου γενικότερα. Πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη και η συμμεταχείριση. Στο πώς ε, αντιμετωπίζουμε το θέμα των μεταναστών και των προσφύγων από την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων, ειδικών των γυναικών και κοριτσιών, επειδή υπάρχουν κάποια σημεία πίεσης όπου συγκεντρώνονται οι άνθρωποι αυτοί. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε κάποιους συγκεκριμένους ειδικότερους τομείς. Πρώτα απ' όλα η σεξουαλική βία. Ένα από τα βασικά σημεία που με απασχόλησαν στη γνωμοδότηση είναι το θέμα της βίας, ιδίως της σεξουαλικής, διότι οι γυναίκες που ετούνται άσυλο είναι ιδιαίτερως ευάλωτες, συχνά είναι μόνες, ε, χωρίς την υπόλοιπη οικογένειά τους και έχω διαβάσει αποτρόπες εκθέσεις ε, για γυναίκες και ε, κορίτσια που έχουν ξεφύγει από συνθήκες πολέμου με πολύ δύσκολα ταξίδια για να ξεφύγουν από τις συνθήκες αυτές, από, περνώντας από Μαρόκο και Λιβύη και θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όσοι προσπαθούν να βοηθήσουν ή ε, τα μέλη των διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων θα τις βοηθήσουν να ξεπεράσουν αυτές τις τραυματικές εμπειρίες. Πολλές μάλιστα μπορεί να μείνουν έγκυες λόγω ε, της σεξουαλικής βίας. Αυτό κάνει την τραγική του ιστορία ακόμα χειρότερη. Δηλαδή να ξεφεύγει, να προσπαθεί κανείς να τραπετεύσει από τον πόλεμο ή τις διώξεις και επιπλέον να πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας και να μένει και έγκυος. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε κατεπηγόντως. Έπειτα υπάρχει το θέμα των εγκαταστάσεων υποδοχής. Πρόσφατα υπήρξε μια έκθεση από ε, αγγλική ε, οργάνωση για τις γυναίκες εργαζομένους εργαζόμενες οι οποίες πολλές φορές έχουν κρατηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από αίτηση ασύλου για πολύ καιρό και έχουν ε, ε, αυτοκτονήσει τελικά. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη ακόμα και στις συνθήκες κάτησής του, οι προηγούμενες τραυματικέ του εμπειρίες. Δεν είναι μόνο το ότι αντιμετωπίζουν στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά το ιστορικό τους γενικότερα. Δηλαδή το ότι έφτασαν σε ένα νέο μέρος, μια νέα χώρα, αντιμετώπισαν όλη τη γραφειοκρατία, τι διοικητικέ δυσκολίε τον πόνο και την ταλαιπωρία από την οποία έχουν περάσει, θα πρέπει λοιπόν το ιστορικό τους προηγουμένως να ληφθεί υπόψη. Δηλαδή να μην τους φερθούν τόσο άσχημα που τελικά να καταλήξουν να αφαιρούν οι ίδιες τη ζωή τους. Ε, το λαθρεμπόριο και η εμπορία είναι ένα επίσης μεγάλο ζήτημα ε, στο τι συμβαίνει στη Μεσόγειο. Ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση, υπάρχουν στενοί συσχετισμοί με την λαθρεμπορία ανθρώπων και οι διακινητές ε, στη θάλασσα πολλές φορές είναι οργανωμένοι σε συμμορίες και οι άνθρωποι που προσπαθούν να δραπετεύσουν είναι θύματά τους. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τους ε, διακινητές αυτούς και θα πρέπει να κάνουμε διάκριση της διακίνησης ανθρώπων από το λαθρεμπόριο. Υπάρχουν δύο διαφορετικά φαινόμενα και από νομικής ε, σκοπιάς και στην πράκτη πράξη. Διότι η διακίνηση, η εμπορία ανθρώπου είναι παραβίαση των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ενώ η λαθρεμπορία ανθρώπων έχει να κάνει με οικονομικά ωφέλη. Θα πρέπει λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε με τον σκοπιμότερο τρόπο. Επίσης υπάρχει και το όλο ζήτημα της εμπορίας ανθρώπου και του λαθρεμπορίου που πρέπει να το κατανοήσουμε καλύτερα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται πολύ καλή δουλειά για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Όμως, όλο ιδιαίτερο αφορά το τι συμβαίνει στη Μεσόγειο και θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να κατανοήσουμε το φαινόμενο. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, το θέμα αυτό είναι άκρο σημαντικό. Θα πρέπει να έχουμε ως Επιτροπή των Γυναικών ε, μια συγκεκριμένη τοποθέτηση μέσα από τη γνωμοδότησή μας. Παρόλο που δεν είναι ευχάριστο το θέμα, οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Και ε, μόλις ε, φτάσει στα χέρια μας και έκθεση ΛΥΜΠΕ θα φροντίσουμε η γνωμοδότησή μας να συμπεριλάβει ή να, συμπεριληφθούν οι δικές μας ιδέες σε εκείνη την έκθεση. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την όλη κατάσταση, είναι και αυτό πολύ σημαντικό, για να μπορούμε να γύρουμε αυτά τα σημαντικά θέματα για τον τρόπο που ε, γυναίκες και τα κορίτσια αντιμετωπίζονται και για να προσπαθήσουμε να προλάβουμε τον πόνο και την ταλαιπωρία που περνούν. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Χάνεμπολ. Η κυρία Μίλναρ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Ειλικρινά θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Χόνιμπολ, τη συντάκτρια γνωμοδότησης για τη γνωμοδότησή της. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αναμφίβολα, και πρέπει να αναγνωρίσουμε και τη διάσταση του φύλου στο φαινόμενο αυτό της μετανάστευσης. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για διαρθρωτικό ζήτημα. Γιατί οι γυναίκε αποτελούν μέρο των μεταναστευτικών αυτών ροών και οδηγούνται σε δύσκολη θέση που τις καταστά περισσότερο ευάλωτε από ότι τους άντρες. Κάτι το οποίο πολύ καλά και με λεπτομέρειες περιγράφει η συντάκτριά μας. Αυτό λοιπόν που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι το εξή. Πρώτον, να σπάσουμε τα στερεότυπα που υπάρχουν για τι μετανάστριε. Δεύτερον, πρέπει να λάβουμε υπόψη μα τη διάσταση του φύλου κάθε φορά που συζητάμε για το άσυλο. Και τρίτον, δεν πρέπει να υποτιμάμε το τι συμβαίνει άπαξ και αρχίσει ή πρέπει να αρχίσει η διαδικασία τη ε, ολοκλήρωση. Πρέπει ένα πράγμα να έχουμε υπόψη μας και αυτό είναι ότι η γυναίκα μετανάστρια ακόμα και αν είναι μορφωμένη θα βρει δουλειά σίγουρα πολύ κατώτερη των προσόντων της, αν το συγκρίνουμε αυτό με τις ντόπιε γυναίκες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κονόσκα έχει τώρα το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, εγώ μιλώ εξ ονόματος της κυρίας Κοράτσα Μπίλτ, που είναι σκιώδη συγγήτρια. Έτσι λοιπόν το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αναγνώσω το κείμενο που μου έχει δώσει. Χαίρομαι λέει για τη γνωμοδότηση για την κατάσταση στην ε, Μεσόγειο, της μετανάστευσης δηλαδή, και για την συνολική αυτή προσέγγιση στα προβλήματα των μεταναστριών. Και ιδίως για το θέμα της άσκησης βίας κατά γυναικών, οι οποίες πέφτουν συχνά θύματα και σεξουαλικής βίας στη διάρκεια του ταξιδιού. Ιδίως πρέπει να προσέξουμε τις έγκυες γυναίκες και τα παιδιά. Ως σκιώδη συγγήτρια έχω ορισμένε προτάσεις και κάποιες τροπολογίες για να φωτίσω ορισμένα πιο σημαντικά σημεία. Θα ήθελα να γίνει πιο συνολική και συνεκτική προσέγγιση, ιδίως στη διακίνηση, στην παράνομη διακίνηση των μεταναστών και μεταναστριών, ιδίω για το θέμα αγνοούμενων ασυνόδευτων ανηλίκων που πέφτουν θύματα κατάχρησης. 50% των ασυνόδευτων παιδιών εξαφανίζονται από τα κέντρα φροντίδας λίγες ώρες μετά από την άφηξή τους εκεί και δεν ξαναβρίσκονται ποτέ. Αυτό κυρίως ε, πλήττει νεαρά κορίτσια τα οποία τελικά εξαναγκάζονται σε πορνεία. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη ανάγκη να καταπολεμηθεί αυτή η παράνομη διακίνηση και να συλληθούν οι διακινητές. Θέλω να γίνει και αναφορά και στα θύματα βίας και στην ε, συνθήκη της Ισταμπούλ, επίσης στις γυναίκες θύματα βιασμών που χρησιμοποιείται ως πολεμικό μέσο να προστατεύονται οι γυναίκες σε ζώνες συγκρούσεων, διότι η πλειοψηφία των προσφύγων είναι πρόσφυγες από αιστείες συγκρούσεων. Έστειλα, ε, μάλιστα, μάλλον ευχαριστώ την εισηγήτρια για την γνωμοδότηση και θα συνεχίσω να συνεργάζομαι και μαζί της και με τους άλλους συνεισηγητές. Eh, Ευχαριστούμε. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο για να κλείσουμε αυτό το θέμα. Η κυρία Χόνεμπολ, για να απαντήσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τους σκιώδεις. Σίγουρα είναι ένα από τα θέματα που θα συνεργαστούμε πολύ καλά όλοι στην Επιτροπή μας. Συμφωνώ με όλα όσα είπατε και θα λάβω υπόψη μου τα όσα αναφέρατε. Νομίζω όλοι είμαστε στην ίδια γραμμή και θα συνεχίσουμε. Ολόκληρη η Επιτροπή μας πρέπει να είναι ενωμένη σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να αρχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράση από αυτού. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε κύριε Χόνιμπολ. Τώρα, πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, η οποία θα λάβει χώρα στις 10 και 4, μας μένει η συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Ο κύριος Ουρτασούν είναι στο δρόμο από ό,τι φαίνεται. Α, όχι, ο κύριος Σεμπαστιά. Εκ μέρους του κύριου Ουρτασούν θα πάρει το λόγο από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, ναι, εκ μέρους του συναδέρφου Ουρτασούν, ο οποίος κάπου έξω από τις Βρυξέλλες έχει μπλοκαριστεί, προσπαθεί να φτάσει. Θα σας παρουσιάσω εγώ την έκθεσή του. Το βασικό θέμα είναι ότι θέλουμε να απαιτήσουμε να συμπεριληφθεί η διάσταση του φύλου στις πολιτικές που έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Δουλεύει σε δύο άξονες. Απ' τη μια είναι επικριτικός και από την άλλη ζητάει αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πολιτικών για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ώστε να δούμε πόσο λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φίλου στις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επικρίσεις. Δυστυχώς πρέπει να πούμε ότι στην στρατηγική Ευρώπη για το 2020 η διάσταση αυτή του φύλου δεν υπάρχει αρκετά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να το κάνει. Απαιτούμε να γίνει. Από την άλλη, οι ειδικέ συστάσεις αναχώρα πρέπει να έχουν συστάσεις για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Υπάρχει μεν στα λόγια, αλλά στην πράξη στις πολιτικές δεν το βλέπουμε. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να απαιτήσει να καλυφθούν τα κενά αυτά. Όσον αφορά τώρα την αξιολόγηση, αυτό που ζητάμε είναι οι χώρες να παρουσιάζουν τα στοιχεία όσον αφορά τα δύο φύλλα για να ξέρουμε πολύ καλά ποιε είναι οι επιπτώσει επί των γυναικών των πολιτικών που εφαρμόζουμε. Αν δεν έχουμε τέτοια στοιχεία αναφύλλω, τότε δεν μπορούμε να ξέρουμε κατά πόσο τηρούνται ή δεν τηρούνται περισσότερο ή λιγότερο οι ε, πολιτικές μας σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων. Έτσι μόνο θα μπορούμε να αξιολογήσουμε τις πολιτικές μας και θα γνωρίζουμε κατά πόσο πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση, κατά πόσο το χάσμα ε, μειώνεται ή αντίθετα αυξάνει ή διατηρείται. Κάτι το οποίο για μας θα ήταν αποτυχία όσον αφορά τις πολιτικές του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αυτές είναι οι προτάσεις πάντως που περιλαμβάνονται στο κείμενο. Περιμένω τώρα την άποψη των συναδέλφων από τις άλλες πολιτικές ομάδες προκειμένου να συμπληρωθεί το κείμενο αυτό. Πάντως η Επιτροπή πρέπει να είναι σαφής. Αν δεν υπάρχει σαφής βούληση από πλευράς του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου να λάβει υπόψη τη διάσταση του φύλου οι επικρίσεις θα συνεχίζονται. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Σεμπαστιά. Είναι σημαντικό πράγματι το ότι η Επιτροπή μας ετοίμασε τη γνωμοδότηση αυτή. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε εξάμεινο πρέπει να αποφαίνεται σχετικά με τις συστάσεις που γίνονται προς τις χώρες μέλη. Το να μην λαμβάνεται υπόψη διάσταση του φύλου, αυτό είναι πολύ αρνητικό. Βεβαίω και επανελειμμένα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στι συστάσεις αυτές η διάσταση του φύλου. Αλλιώς είναι παράληψη που δεν δικαιολογείται. Σας ευχαριστώ λοιπόν που αναλάβατε την πρωτοβουλία αυτή για τέτοια γνωμοδότηση ελπίζω στην Επιτροπή επί να ληφθεί υπόψη, η απόψή μας. Τώρα, παρεμβάσεις. Ποιος θέλει το λόγο? Φαίνεται ότι έχουμε μπει κάπως σε κλίμα διακοπών. Ότι λίγο, λίγο, σιγά σιγά έχουμε κουραστεί, όλοι περιμένουμε τις διακοπές. Εντάξει, είναι λογικό. Και το κλίμα αυτό το βλέπουμε και εδώ στις συζητήσεις μας, γι' αυτό δεν είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να πάρουν το λόγο. Η κύριε Κολόσκο, όμως, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ολόκληρη σειρά εκθέσεων έχουμε εδώ και έχω και εγώ να πω κάτι ειδικά για την έκθεση που έχουμε μπροστά μας. Αφού πρώτα ευχαριστήσω για την εργασία του εισηγητού αλλά και για το έγγραφο αφού το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο είναι το βασικό εργαλείο συντονισμού για την επίτευξη των στόχων του 2020. αποτελεί και την βάση για τις εθνικές οικονομικές πολιτικές και για τη συνοχή στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν σημαντικό να οικοδομηθεί σωστά και συνεκτικά. Αυτό το 75% της απασχόλησης στην Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν επιτύχουμε την σωστή σύνδεση μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Και αυτό ισχύει ιδίω για τι γυναίκε. Και αυτό ισχύει επίση ιδίω για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο για την προσπάθεια επίλυση των προβλημάτων και καλύψη των κενών. Οι τροπολογίες θα μα επιτρέψουν, ελπίζω, να εμβαθύνουμε στη συζήτηση αυτή και όπω είπα το θέμα είναι η ισότητα μέσα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ζητά κανένα άλλο το λόγο από ό,τι βλέπω. Ο κύριος Σουρτασούν έφτασε και έχουμε ακόμα 10 λεπτά πριν ε, την ώρα των ψηφοφοριών. Ο κύριος Σουρτασούν έχει το λόγο για να συμπληρώσει τόσα είπε ο συναδελφός του, ο κύριος Σεβαστιά, που πολύ καλά μας εξήγησε. Καλά, θα είναι δύσκολο, δεν ήμουν εδώ, ποτέ, δεν ξέρω τι είπε. Ζητώ συγγνώμη. Είχε φοβερή κίνηση στις Βρυξέλλες, γι' αυτό δεν μπόρεσα να φτάσω στην ώρα μου. Το μόνο που θέλω να σας πω, έχω δει το κείμενο βέβαια αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να συμπεριληφθούν τα θέματα που πιστεύουμε ότι είναι σημαντικά μέσα στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Σίγουρα ο συνάδελφος σας τα είπε. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι τόσο η αναχώραση στάσης όσο οι μεταρρυθμίσεις των χωρών πρέπει να αξιολογούνται όσον αφορά τη διάσταση του φύλου. Επίσης η γνωμοδότηση, κάτι άλλο σημαντικό που λέει, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι που θεωρούμε εμεί σημαντικό. Με τις διάφορες μεταρρυθμίσεις που γίνονται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιπτώσεις που έχουν όλα αυτά πάνω στη διάσταση του φύλου. Επίσης, ξέρετε ότι γίνεται σημαντική συζήτηση αυτή την εποχή στην διαδικασία για τις μακροοικονομικές ε, ανισορροπίες, κατά πόσο πρέπει να συμπεριληφθούν κοινωνικοί δείκτες ή όχι, είναι ο αγώνας που δίνει η κυρία Τάισεν. Εμείς συμφωνούμε να υπάρχουν κοινωνικοί δείκτες και δείκτες που να συμπεριλαμβάνουν τη διάσταση του φύλου. Είναι ζωτική σημασία. Το λέμε στη γνωμοδότησή μας. Τέλος, υπάρχει και ο προβληματισμός στο κείμενο για τις επιπτώσεις που θα έχει το πρόγραμμα Juncker, οι επενδύσεις, το επενδυτικό πακέτο Juncker στη διάσταση του φύλου. Και εδώ μερικοί τομείς επηρεάζουν άμεσα την ισότητα των δύο φύλων. Γι' αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και εκεί. Θα έχω επαναλάβει δίχως άλλο διάφορα που είπε ο συνάδελφος Σεμπαστιά, δεν θέλω να συνεχίσω. Να επενθυμίσω μόνο ότι η προθεσμία είναι πολύ στενή, είναι τώρα την Παρασκευή. Ελπίζω λοιπόν μέχρι την Παρασκευή να έχω τις ε, τροπολογίες σας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Ουρτασούν. Όσον αφορά το τελευταίο που είπατε, ακριβώς θα σας έλεγα ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και για την κυρία Χόνεμπολ και για τη δικιά σας ε, έκθεση. Λοιπόν, υποβολή τροπολογιών για την έκθεση αυτή όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμενο είναι 17 Ιουλίου. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα λάβει χώρες 15 Σεπτεμβρίου. Θα ψηφίσουν στην Επιτροπή ε, Οικονομικός 13 Οκτωβρίου και τον Οκτώβριο θα ψηφίσουμε και στην Ολομέλεια. Και έρχομαι τώρα στην έκθεση Honeyball για την Μεσόγειο. Εδώ, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 8η Σεπτεμβρίου. Ψηφίζουμε εδώ στις 15 Οκτωβρίου, στη Λίμπε 16 Νοεμβρίου και στην Ολομέλεια το Δεκέμβριο. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τις συζητήσεις για τις εκθέσεις. Σας κάνουμε 5 λεπτά ένα μικρό διάλειμμα, διακοπή μέχρι να πάει 10 και 4 γιατί ίσως κάποιοι συνάδελφοι να φτάσουν ακριβώς στις και 4 για τις ψηφοφορίες. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας αρχίσουμε με την ψηφοφορία, παρακαλώ. Comenzamos con los votos, eh, espero. Ας αρχίσουμε. Φαντάζομαι ότι έχετε όλοι τις κάρτες σας, τις κάρτες για την ψηφοφορία, έτσι γιατί θα τις χρειαστούμε κάποια στιγμή. Αρχίζουμε λοιπόν τις ψηφοφορίες με την ψηφοφορία της έκθεσης της κυρίας Βόζαμπεργκ. Σήμερα είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για την ε, κατάσταση των γυναικών στον επιστημονικό και πανεπιστημιακό χώρο και για τους όρατους φραγμούς που αυτές αντιμετωπίζουν. Τροπολογία αριθμό 40. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα ελέγξουμε καλύτερα. Τροπολογία 43. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 53 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 54 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63, 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 67 κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Δεν ψηφίσαμε την 63 μου λένε. Πρέπει να ψηφίσουμε την 63. Τροπολογία 63 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68 τώρα υπέρ. Κατά. Τι. Τι ψηφίσαμε λέει η πρόεδρος. Α. 69 λοιπόν τότε. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική, α όχι δεν είναι συμβαστική, είναι μια προφορική τροπολογία του κυρίου Σεμπαστιά. Παρακαλώ. Ή αν τη γνωρίζετε να τη ψηφίσουμε. Την έχετε, την έχετε, έτσι δεν είναι. Ωραία, ψηφίζουμε την προφορική τροπολογία του κ. Σεμπαστιά. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 71. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 72. Υπέρ, κατά, Αποχές θα ελέγξουμε. Τροπολογία 72. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 73 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 78 ήταν. Αυτό είπα. Δεν είπα αυτό. Ωραία. Θα αναλάβω εγώ την ευθύνη. Δεν θα τα βάλουμε με τις διερμηνείς τώρα, λέει πρόεδρος. 78, πάση περιπτώσει. 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 79. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 84 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 97 έχει αποσυρθεί. 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 103 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 105 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 3 του κ. Σεβαστιά υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 108 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 114 λέει πρόεδρος. Α, 113 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 4. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Θα ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 4. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά, Αποχές. Απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία αριθμός 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία αριθμός 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία της έκθεσης με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η έκθεση, 30 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά. Συγχαρητήρια κυρία Βόιζαμπεργκ. Και περνάμε τώρα στην επόμενη ψηφοφορία που είναι για το Γενικό Προϋπολογισμό του 2016 say you know, or uh, in the first moment I said that we have to do that. Okay. Uh, one, two. Ah, okay. Πασάμε στα la Θα περάσουμε στην ψηφοφορία επί των τροπολογιών. Πώς τις έχετε εδώ, 6.000, 6.000 λοιπόν ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6.001 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 6.030 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτή. 6.002 νέα, νέα θέση του Συμβουλίου υπέρ κατά αποχές δεν βλέπω να σηκώνετε τα χέρια ας ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά 6.002 Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται λοιπόν. 6.003 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6.004 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται και αυτή. 60.05 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6006 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6007 επίσης νέα διατύπωση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6024 νέα βερσιόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 6008 νέα εκδοχή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6009 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6025 νέα διατύπωση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6029 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6.031 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 6.032 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 6.027 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 6.010 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 6.011 νέα διατύπωση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6.012 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 6.013 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6.028 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6.014 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6.015 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6.020 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6.021 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6.022 νέα διατύπωση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6.023 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6.016 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6.019 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6.017 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το υπόλοιπο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6.026 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και 6.018 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εγκρίθηκαν λοιπόν οι τροπολογίες. Περνούμε στο επόμενο, στην επόμενη έκθεση. Γνωμοδότηση για την πολιτική συνοχής Enmienda de compromiso. Uy, no. La 21. Votos a favor. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39. Με μια γλωσσική διόρθωση. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεν είναι σαφές θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά το δεύτερο τμήμα της 39. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για τα 49. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 50 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε τις ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 51. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε τώρα τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 21 ψήφοι υπέρ, 1 κατά και 9 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Ρουτασούν. Ψηφίζουμε τώρα την έκθεση όσον αφορά το στρατηγικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για την περίοδο 2014-2020. Η κυρία Μπορσάν είναι η, η συντάκτρια γνωμοδότησης. Τροπολογία 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 33. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ωραία, για την 35. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε για την τροπολογία 39. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές Εγκρίνεται νομίζω, αλλά προτιμώ να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Συμβαστική 2. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας. Καλά το είδα. Αλλά βέβαια δεν είχα πιστοσύνη στον εαυτό μου. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 48 τώρα. Έτσι δεν είναι. Ναι. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 49. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Α, τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42 λέει πρώτος, 52 προφανώς. Κατά τμήμα πρώτο τμήμα υπέρ. 52 διορθώνει τώρα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 53. Υπέρ. Να ελέγξουμε ποιο, το δεύτερο τμήμα. Είπα ότι απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε δεύτερο τμήμα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη φοφορίας.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 εγκρίνεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 77 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4 υπέρ,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 θα ελέγξουμε εδώ. Τροπολογία 13. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Θα ελέγξουμε για την τροπολογία 24 παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρας της Καθόλου καλά δεν το είχα δει. Προφανώς εγκρίνεται. 25 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές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 Σε Πέρα τη οφορίες. Εγκρίθηκε 19 ψήφοι υπέρ, 4 κατά και 8 αποχές. Συγχαρητήρια κύριε Μπόρσαν. Ψηφίζουμε τώρα την έκθεση για τη διάσταση του φύλου. Πρόκειται για την ε, υλοποίηση των μικροχρηματοδοτήσεων. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Με προφορική τροπολογία του κύριου Ορτασούν που θέλει και το λόγο. Πρέπει να σας εξηγήσω λίγο την προφορική τροπολογία γιατί δεν την έχετε. Λέτε εξή. Αλλάζει τροπολογία θα λέτε εξή. Εφόσον όλο και μεγαλύτερο αριθμό γυναικών που συμμετέχουν στην αγορά εργασία είναι αυτέ που τρέφουν την οικογένειά του. Αυτή είναι η αλλαγή που ζητάμε σε σχέση με το αρχικό. Ωραία, συμφωνούμε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 των τροπολογιών για τη διάσταση του φύλου όσον αφορά την έκθεση της κυρίας Λεγκρίπ. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συνεπώς, εδώ ολοκληρώθηκαν οι ψηφοφορίες. Τελειώσαμε ακριβώς την ώρα μας. Όπως προβλεπόταν. Μπράβο. Παρά την προεδρό σας, η οποία έχει μπερδευτεί λίγο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Τώρα, περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την Λουξεμβουριανή Προεδρία. Yeah,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 Συνεχίζουμε. Τώρα θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την Λουξεμβουριανή Προεδρία. Να αρχίζει αυτό το μήνα. Οπότε καλωσορίζουμε εδώ την κυρία Μούτς, που είναι Υπουργός Ίσων Ευκαιριών Συνηθίζουμε στην Επιτροπή μας να προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε και να προβάλλουμε θέματα τα οποία για μας αποτελούν προτεραιότητα στα πλαίσια των εργασιών των διαφόρων προεδριών του Συμβουλίου. Επιθυμία μας λοιπόν είναι η συνεργασία αυτή να γίνει ακόμα πιο στενή μέσα στους επόμενους μήνες με τη Λουξεμβουριανή Προεδρία. Υπάρχουν ζητήματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη και τα οποία ελπίζουμε να προωθήσει η Λουψεβουριανή Προεδρία. Να προωθήσει τέτοια σχέδια και προγράμματα. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μούτς και μετά θα συζητήσουμε με τους συντονιστές των διάφορων πολιτικών ομάδων. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Λοιπόν, θέλω να νιώσετε ότι βρίσκεστε σε ένα χώρο που θέλει συνεργασία μαζί σας και σας ευχόμαστε καθημερινά θετικά αποτελέσματα για το καλό της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας στόχος τον οποίο συμμεριζόμαστε όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Σενιώρα Πρεζιντέντε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Με μεγάλη χαρά θα σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας στην ομιλία μου θα αναφέρω όχι μόνο τις προτεραιότητες της Προεδρίας μας, αλλά θα τοποθετηθώ και σε σχέση με την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, που εξ όσων καταλαβαίνω σας ενδιαφέρει ιδιαίτερος. Η Λουξεμβουργιανή Προεδρία ξεκινά σε μία περίοδο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις. Μιλάμε για κρίση. Οι άντρες και οι γυναίκες δεν είναι ίσιος προς την κρίση και τις συνεπιές της. Τα μέτρα λιτότητας που αποφασίστηκαν σε πολλές χώρες έχουν πλήξει ιδιαίτερως τις γυναίκες γιατί είναι πιο εκτεθειμένες στην επισφάλεια των συνδικών εργασίας, την απώλεια, απολύσεις, την φτώχεια, την κοινωνική υποβάθμιση. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τις γυναίκες που έχουν να αντιμετωπίσουν ε, πολλαπλά προβλήματα όπως οι μόνες μητέρες, οι νέες ή αυτές που προέρχονται από εθνικές, εθνοτικές μειονότητες. Είναι προβλήματα που εντείνονται ακόμη περισσότερο σε περίοδους κρίσης. Μια από τις πολιτικές λοιπόν της Ένωσης είναι να εντοπίσουμε τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών για να διασφαλίσουμε ότι κάθε στρατηγική καταρτίζεται για να αντιμετωπίσει την κρίση και να αναθερμάνει την οικονομία αντιμετωπίζοντας τις δυσμενείς επιπτώσεις στους άνδρες και όλος ιδιαίτερα στις γυναίκες. Το Σεπτέμβριο του 2014 η έννοια του gender budgeting, δηλαδή του προπολογισμού βάση των αναγκών των φύλων, αποτέλεσε το εργαστήριο ε, το θέμα ενός εργαστηρίου με αντικείμενο τις προτεραιότητες για το θέμα αυτό μετά το 2015 και οργανωμένο από τις ε, ανώτερες αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω οι προτεραιότητες για το gender budgeting δείχνουν τι σημασία έχει το πεδίο αυτό που πρέπει να εξερευνηθεί για να δούμε τις διαφορετικές επιπτώσεις της δημοσιονομικής πολιτικής και πώς ε, αυτή έχει συνέπειε διαφορετικέ για του άντρε και τι γυναίκε. Υπάρχουν συστάσει ιδιαίτερα επικοδομητικέ από αυτό το εργαστήριο, όπω τα παραδείγματα καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε κάποια κάτι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία μα παροτρύνουν να ανατρέξουμε περισσότερο στην τεχνογνωσία που διατίθεται και που ε, και που ε, μας διαθέτουν κάποιοι φορείς όπως το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ισότητα των Φύλων. Η στρατηγική για την ισότητα των φίλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ολοκληρώνεται φέτος και στα μάτια της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας η δυνατότητα να μπορέσουμε να σωματώσουμε την πολιτική της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε άλλες στρατηγικές είναι κατά την άποψή μου ένα ψευδές ε, σήμα και αντίθετο στο ρεύμα της πορείας που έχουμε ακολουθήσει ως τώρα για να αντιμετωπίσουμε ε, ε, τον αντίκτυπο της κρίσης. Θα πρέπει να δούμε την εμβέλεια των προβλημάτων που σχετίζονται με την ανισότητα ανδρών και γυναικών σε πολλούς τομείς που θα πρέπει να μας απασχολήσουν η αρχή του gender mainstreaming, της ευθυγράμμισης των ε, αναγκών των δύο φύλων πρέπει να ενσωματωθεί σε κάθε πτυχή της πολιτικής, γιατί η έννοια του φύλου είναι και αναγκαία ως προς την προβολή και την κατανόηση της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα πρέπει να είναι ξεχωριστή και θα επιτρέπει να εντοπίσουμε τα αίτια των ανισοτήτων μεταξύ και γυναικών σε όλους τους πολιτικούς τομείς και έπειτα να προτείνουμε συγκεκριμένους στόχους και μέσα για να πετύχουμε τους στόχους μας και να υπάρχει πραγματική ισότητα μεταξύ των φύλων. Αλλά το Λουξεμβούργο το σέλος θα δεσμευτεί προς αυτή την κατεύθυνση, γι' αυτό και συνείδησα την υπεύθυνη επίτροπο για να την ευαισθητοποιήσω ως προς το θέμα αυτό και ε, συνυπογράψαμε επιστολή από 21 κράτη-μέλη που το απευθύναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εμείνουμε στην ανάγκη να διατηρήσουμε ακριβώς την κοινοτική στρατηγική που θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Κοινοτική στρατηγική για την ισότητα. Πίεση λοιπόν για να υπάρξει μεγαλύτερη προβολή, αλλά και θέμα προτεραιοτήτων και πολιτικής αξιοπιστίας. Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου θεωρεί το θέμα της ισότητας ανδρών και γυναικών ως θέμα προτεραιότητας ως προς την εθνική δράση αλλά και την διεθνή. Γι' αυτό η νέα κυβέρνηση θέσπισε τον ε, Δεκέμβριο του 2013 την ισότητα ανδρών και γυναικών ως ε, κατευθυντήρια αρχή της κυβερνητικής ατζέντα. Είμαστε μια από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που έχει ιδρύσει εντελώ αυτόνομο Υπουργείο που ασχολείται με την ισότητα ανδρών και γυναικών από το 1995. Και αυτή η διάθεση να επιτελέσουμε πρόοδο στην ισότητα μεταξύ άντρων και γυναικών αντικατοπτρίζεται κυρίως στο τρίτο μας πρόγραμμα δράσης, το οποίο εγκρίθηκε από τη νέα κυβέρνηση, προκειμένου να τεκμεριωθεί η συλλογική υπευθυνότητα της κυβέρνησης για τα θέματα αυτά, πέραν του προγράμματος δράση για την ισότητα, Συζητήσαμε με όλα τα άλλα Υπουργεία για να ε, ορίσουμε τους πολιτικούς μας στόχους και να επιδιώξουμε από κοινού την υλοποίησή τους. Γι' αυτό η ευθύνη μας είναι συλλογική και διυπουργική. Κάθε λοιπόν υπηρεσία εντόπισε συγκεκριμένους στόχους προς επίτευξη για τα ερχόμενα χρόνια σε αυτό το πνεύμα συνεργασίας και δι-υπουργική συνεργασίας το Υπουργείο Ισότητας των Ευκαιριών θέλει να προωθήσει την ίδια μορφή ισότητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου είναι θέματα που απαιτούν μία διατομεακή προσέγγιση με κοινέ προσπάθειες σε όλους τους πολιτικούς τομείς και το ίδιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατά την Ιταλική Προεδρία, πιο συγκεκριμένα τη στιγμή της διάσκεψης για την ισότητα των φίλων στην Ευρώπη, Unfinished Business, ατελείωτη ε, πορεία στη Ρώμη, η Λετωνία και το Λουξεμβούργο με τι τριπλές προεδρίες ε, συνεπέγραψαν μια δήλωση για να προωθήσουν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η κοινή αυτή δήλωση ορίζει από τη μια τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη δράση μας και μετά την πολιτική, ε, τις πολιτικές των τριών προεδριών. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται τα διάφορα στοιχεία της πολιτικής ισότητας ανδρών και γυναικών ε, και που έρχονται να εκτελεστούν στο εξάμενο της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας. Πρώτη προτεραιότητα, η ισορροπή συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην διαδικασία λήψη αποφάσεων, οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων. Δεδομένου ότι αυτή παραμένει μια μεγάλη αδυναμία στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει ανάγκη να δράσουμε περισσότερο για την ισότητα ανδρών και γυναικών στη διαδικασία λήψης πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τους αριθμούς που πρόσφατα δημοσιεύτηκαν Ε, βάσει του δίκτυ ισότητας ε, των δύο φύλων που όλοι γνωρίζουμε ως προς την λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι άντρε ε, κατέχουν τρία τέταρτα των υπουργικών θέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και αν υπάρχουν σοβαρές αποκλήσεις μεταξύ των διαφορών χωρών. Η εικόνα είναι παρόμοια προς την εκπροσώπηση των γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια όπου βέβαια έχουν επιτευχθεί κάποιες σχετικές πρόοδοι χωρίς όμως να μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιο άλμα πρόοδου, το οποίο ουσιαστικά θα επιθυμούσαμε. Η κατάσταση είναι καλύτερη σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, όμως η αναλογία είναι 1 τρίτο προς 2 τρίτα υπέρ των ανδρών φυσικά. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία λήψη αποφάσεων σε θέματα οικονομίας, εν γέννη συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια όλος ο φτάνει το 16% κατά μέσο όρο. Κάτι που είναι μάλλον ένα πολύ μέτριο αποτέλεσμα, ακόμη και αν υπάρχει μια σχετική βελτίωση 6% σε σχέση με το 2005. Το 2012 μόνο 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφταξαν σε ίσο ποσοστό, του 16% δηλαδή, ή ξεπέρασαν το 20%. Οι αριθμοί είναι σαφείς. Δείχνουν ότι πρέπει να ενισχύσουμε όλες τις εθνικές μας προσπάθειες, αλλά και τις διεθνείς, για να έχουμε περισσότερες γυναίκες στην πολιτική πολιτική αρένα και στην, στο οικονομικό πεδίο. Η Προεδρία μας λοιπόν δεν θα αφιστεί προσπαθειών για να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Επίσης οι πολιτικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου ε, είναι μεταξύ άλλων να φτάσουμε στο 40% της εκπροσώπησης στα υψηλά κλιμάκια στους τομείς των δημόσιων υπηρεσιών στο 2019. Για, τις, ε, ε, για τον ιδιωτικό τομέα η κυβέρνηση στηρίζει την πρόταση Ευρωπαϊκής Οδηγιά της Ποσοστώσης Βάσης Νομοθεσίας για τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείε και ταυτόχρονα πρόκειται να εντείνω το πρόγραμμα για τις θετικές ενέργειες που θα επιτρέπουν στις ιδιωτικές επιχειρήσεις να επιταχύνουν την υλοποίηση και την επιδίωξη της καλύτερης εξισορρόπησης. Στο Λουξεμβούργο η εκπροσώπηση των γυναικών για την διαδικασία λήψη πολιτικών αποφάσεων ξεπερνά λίγο το ποσοστό ε, του σκέλου των οικονομικών αποφάσεων, αλλά παραμένουν λιγότερε από του άντρε. Η κυβέρνηση έχει την πρόθεση ε, εφ' να, μεταβάλει, να προσαρμόσει την νομοθεσία ως προς το θέμα αυτό για να φτάσουμε στο 40% της ε, προσώπησης των ε, δύο φύλων, των γυναικών δηλαδή, στα ψηφοδέλτια στις επόμενες εκλογές το 2018. Επίσης ένα βαθμιαίο σύστημα κυρώσεων για μη σεβασμό των ποσοστώσεων είναι κάτι που επίσης προτείνεται κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Θέλουμε να ε, συζητήσουμε το θέμα της συμμετοχής στη διαδικασία λήψης οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων σε κοινοτικό επίπεδο και αυτό να γίνει πρώτη μας προτεραιότητα για τα θέματα ισότητας ανδρών και γυναικών. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι η ενεργός στήριξη για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καλύτερη εξισορρόπηση της εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στους ε, ε, διοικητές, ε, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιριών που είναι εισηγμένε στο χρηματιστήριο από την αρχή της θητείας μου. Έχω εκφράσει τη στήριξή μου για το εγχείρημα της οδηγίας αυτής μέσω διμερών επαφών, επανειλημμένων, συνομιλιών, μια πυκνή επικοινωνίας με πολλούς συναδέλφους και ως προς αυτό το θέμα είχαμε συχνή συνεργασία με την Ιταλική Προεδρία για να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Ήθιστε η Προεδρία του δεύτερου εξαμήνου να αναλύει όσα έχουν πραγματοποιήσει τα κρατη για την υλοποίηση κρίσιμων τομέων τη πλατφόρμας του Πεκίνου προκειμένου να βεβαιωθεί ότι υπάρχει συνέπεια. Η Λουξεμβουργιανή Προεδρία επέλεξε τον τομέα οι γυναίκες στη λήψη αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ισότητα των Φύλων συντάσσει μετά από ε, παραγγελία του Λουξεμβούργου έκθεση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στον τομέα της δήλωσης και του προγράμματος δράσης του Πεκίνου ε, γυναίκες στη διαδικασία λήψη αποφάσεων και στην εξουσία. Τα απορίσματα θα παρουσιαστούν σε μία συνεδρίαση της ομάδας υψηλού επίπεδου για την ευθυγράμμιση των αναγκών των φύλων το Σεπτέμβριο του 2016. Επίσης, σε μια διεθνή διάσκεψη για το θέμα της ισότητας στη διαδικασία λήψης οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων που θα διοργανώσουμε στις 15 και 16 Οκτωβρίου με την ε, επιβεβαιωμένη συμμετοχή του Γερμανού Υπουργού Δικαιοσύνης και της ε, κυρίας Ρέγνερ ε, που είναι ευρωβουλευτής από την Αυστρία και η συγγήτρια για την έκθεση επί του θέματος αυτού. Στην άτυπη σύνοδο του ε, Συμβουλίου Οικονομικών, Κοινωνικών μάλλον, Υποθέσεων ε, την πιο πρόσφατη σύνοδο ε, ελήφθησαν σχετικές αποφάσεις βάσει της έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος. Έπειτα η αγορά εργασίας και η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε αυτήν. Το Λουξεμβούργο στηρίζει την πρωτοβουλία Ευρώπη 2020 ώστε να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης σε 75% στο 2020 οι γυναίκες είναι ένα εργατικό δυναμικό δυνάμει που θα μπορούσε να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει τους στόχους της σχετικά προκειμένου να υπάρξει αυξημένη συμμετοχή των γυναικών την στο χώρο της εργασίας. Και αυτό θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους μας περί απασχόλησης και να υπάρξει κοινωνική ενσωμάτωση αλλά και καταπολέμηση της φτώχειας. Η συνάδελφος θα αναπτύξει περισσότερο το θέμα αυτό στη συνέχεια. Οι αμοιβέ της εργασίας με τρόπο ισότιμο μεταξύ άντρων και γυναικών είναι μια προτεραιότητα θεμελιώδης σημασίας. Όμως, με την δικαιολογημένη πολιτική βούληση να αυξήσουμε το ποσοστό εργασίας των ε, γυναικών και να αυξηθεί η παρουσία των γυναικών στα κλιμάκια και τα αξιώματα ευθύνη είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολήσει από τη σκοπιά της ισότητας και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό το Υπουργείο Ισότητας των Ευκαιριών στο Λουξεμβούργο θα συζητεί το θέμα της κατανομής ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών στον επαγγελματικό και ιδιωτικό βίο. Θα εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να συζητήσουμε στην άτυπη σύνοδο του Συμβουλίου Κοινωνικών Υποθέσεων στις 16 και 17 Ιουλίου, σε λίγες μέρες δηλαδή, και θα δείξουμε έξι πόσο μας ενδιαφέρει η πολιτική ισότητα ε, των φύλων και των ευκαιριών. Όλοι οι υπουργοί απασχόλησης και ίσων ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όπως και κλειμένοι σε αυτή τη σύνοδο. Επιτρέψτε μου να εμβαθύνω λίγο στην προσέγγιση που έχουμε επιλέξει. Οι άνδρες μπορεί και αυτοί να είναι θύματα δικαιωτικής μεταχείρισης ή άνησης μεταχείρισης. Κάτι που έχει να κάνει με τα στερεότυπα και την οτροπία σχετικά με αυτά. Τους ε, κοινωνικοψυχολογικούς ρόλους όπως γίνονται αντιληπτοί τα στερεότυπα αυτά δυσκολεύουν ε, το να αλλάξουν οι παραδοσιακοί ρόλοι που αποδίδονται στους άντρες και τις γυναίκες, ιδίως στο πλαίσιο του συνδυασμού επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για τους άντρες. Άντρες οι οποίοι θα θέλουν να είναι πιο ευέλικτοι για να μπορέσουν να συνδυάσουν τα δύο. Ωστόσο, Υπάρχουν δυσκολίες των παραδοσιακών ρόλων που συνήθως αποδίδονται από την κοινωνία στους άντρες. Είναι αυτοί οι στυλοβάρτες της οικογένειας. Και από την άλλη στις επιχειρήσεις δεν έχει αλλάξει επαρκώς η ώστε να υπάρχει ίδια ευελιξία για τις γυναίκες και τους άντρες για τους άντρες που θέλουν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στον ιδιωτικό τους βίο. Για να είμαστε σαφείς, δεν θέλουμε να βρούμε αμέσως απαντήσεις ή λύσεις ή όλα να αμφισβητηθούν ως προς την πολιτική ισότητα ανδρών και γυναικών, αλλά θέλουμε να ετοιμάσουμε το έδαφος για να μπορέσουμε να μελετήσουμε το θέμα στη διάρκεια των ερχόμενων προεδριών και να μπορέσουμε να δηλήσουμε στοιχεία από τα κράτη-μέλη για να δούμε αν έχουν αναλάβει μέτρα ή έχουν προβλέψει ενέργειες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν παραδείγματα καλών πρακτικών. Θέλουμε να ασχοληθούμε με τρεις μεγάλες ευκαιρίες στο πλαίσιο της άτυπης συνόδου του Συμβουλίου Κοινωνικών Υποθέσεων για να μπορέσουν οι Υπουργοί Απασχόλησης να έχουν συμμετοχή στο όλο θέμα αυτό, να διοργανώσουμε μια πλατφόρμα συναντήσεων στο Υπουργείο που ασχολείται με την ε, ισότητα ε, μεταξύ των δύο φύλων και μετά να καταρτήσουμε ένα κατάλληλο εγώ με θέματα για το ρόλο των ανδρών στην πολιτική τη ισότητα ευκαιριών, στην αγορά εργασία και τη διαδικασία λήψη αποφάσεων πολιτικών και οικονομικών. Θα ήθελα σε αυτό το πλαίσιο να σα ενημερώσω και για μία ακόμη διάσκεψη που θα οργανωθεί κατά τη διάρκεια της Λουξεμβουριανής Προεδρίας, μία διάσκεψη η οποία θα διοργανωθεί από το Υπουργείο ε, Εργασίας και Απασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας και η οποία θα αφορά την ε, ε, ατομική φορολόγηση και την απασχόληση. Η διάσκεψη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των συζητήσεων που μόλις ξεκινούμε και θα πρέπει να γίνουν διυπουργικέ και διεπιστημονικέ προσπάθειε ώστε να προσεγγίσουμε το θέμα τη ισότητα ανδρών και γυναικών από την πλευρά των πολιτικών οικονομία, εργασία, απασχόληση ε, και τη κοινωνική πρόνοια ή τη ε, οικογένεια. Τρίτη προτεραιότητα τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία είναι ότι θέλουμε να προωθήσουμε την αρχή του gender mainstreaming, τη ευθυγράμμιση των αναγκών των φίλων, στι διάφορε πολιτικέ και του οργανισμού ή ιδρύματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω ήδη αναφέρθηκε. Η συνεδρία, η σύνοδος του, ε, άτυπη σύνοδος των Υπουργών ε, ΕΠΣΚΟ στις 17 Ιουλίου θα συζητήσει και το θέμα αυτό. Πρέπει όμως και οι άλλοι σχηματισμοί στο επίπεδο του Συμβουλίου να ασχοληθούν με την προοπτική της ισότητας των φίλων στις εργασίες τους. Ένα παράδειγμα, το πρόγραμμα της κυβέρνησης του Λουξεμβούργου για το εξάμεινο της Προεδρίας μας προβλέπει να ληφθεί υπόψη το θέμα αυτό στον τομέα της έρευνας μία από τις βασικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Θα εμβαθύνουμε στο θέμα αυτό και θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην διάσταση ε, των προσλήψεων βάσει διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής που να είναι διαφανής και χωρίς διακριτική μεταχείριση. Ε, εξασφαλίζοντας έτσι μια καλύτερη παρακολούθηση των θεσμικών αλλαγών σε θέματα ισότητας των φύλων. Τέλος, Τέταρτη προτεραιότητα. Το Λουξεμβούργο θα προβάλλει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει την ισότητα ευκαιριών και δικαιωμάτων των γενικών παντού στον κόσμο. Και μάλιστα βάσει των συστάσεων της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου. Αυτό ισχύει όλος ιδιαίτερο σε θέματα πολιτικών συνεργασίας για την ανάπτυξη και τον ορισμό νέων στόχων για τη χιλιετία, μετά το 2015. Είναι κρίσιμη σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δεσμεύσει, ώστε η ισότητα φύλων, των φύλων, δηλαδή των ανδρών και των γυναικών, να ενσωματωθεί ω διατομιακή προτεραιότητα και ω ε, ξεχωριστός στόχος. Το Μεγάλο Δουκάτο έχει καταβάλει εντατικέ προσπάθειε ω προ την αναπτυξιακή συνεργασία από τότε που ξεκίνησε η εθνική μα στρατηγική για τη συνεργασία και την ανάπτυξη ή την ανθρωπιστική δράση και το Λουξεμβουριανό Υπουργείο για την ε, Αναπτυξιακή Συνεργασία έχει σχεδιάσει και καταρτήσει μια τομεακή στρατηγική για τα φύλλα με στατηγικούς δείκτες και στόχους ώστε να καταμετρούμε τον αντίκτυπο της αναπτυξιακής συνεργασίας για τους άνδρες και τις γυναίκες ξεχωριστά. Στο εθνικό πλαίσιο της πολιτικής ισότητας ανδρών και γυναικών αυτή η προσέγγιση είναι νομίζω υποδειγματική ως προς το ενσωματώνουμε την ευθυγράμμιση των αναγκών των φίλων στις πολιτικές μας. Κυρίες και κύριοι, Έχω πλήρη συνέστηση του γεγονότος ότι ορισμένα θέματα που σας απασχολούν συστηματικά και σας είναι ιδιαίτερα προσφυλή δεν θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια τη προεδρία μα. Κάθε προεδρία πρέπει να εντοπίζει κάποια θέματα προτεραιότητα για αυτό το σύντομο διάστημα των έξι μηνών που αναλαμβάνει καθήκοντα, με κοινέ ευθύνε, συλλογικέ ευθύνε από το τρίο των προεδριών που πρέπει να παρουσιάζουν ένα ποικίλο πρόγραμμα και να αντιμετωπίζουν από κοινού τα θέματα που έχουν οριστεί. Η καταπολέμηση της των μορφών βίας κατά των γυναικών δεν είναι από τα θέματα προτεραιότητας της Προεδρίας μας. Όμως η καταπολέμηση της βίας είναι προτεραιότητα σε καθημερινό επίπεδο για όλους μας. Σας παραπέμπω στην κοινή δήλωση του Τριγώνου Προεδριών που δήλωσε με σαφήνεια ότι οι ανισότητες ανδρών και γυναικών αποτελούν μια παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ότι πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για να εκριζωθούν ε, μεταξύ άλλων οι μορφές βίας που διαπράττονται κατά των γυναικών. Το Λουξεμβούργο συνάδει πλήρως με αυτή την έκφραση και θέλει να αναλάβει δράση κατά της βίας λόγω του φύλου τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε διεθνές. Η χώρα μου διαθέτει μια αποτελεσματική ε, νομοθεσία για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας από το νόμο που ήδη έχει ε, αναθεωρηθεί από το 1993 με μορφές συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών του χώρου αυτού και για να καταμετρηθούν οι διαστάσεις του φαινομένου αυτού στη χώρα μας. Το αρμόδιο Υπουργείο διαρκώς οργανώνει εκστατείες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την πρόληψη αυτών των φαινομένων. Ως τώρα, 36 χώρες της Ευρώπης μεταξύ των οποίων το Λουξεμβούργο, έχουν συνυπογράψει και κυρώσει τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη για την πρόληψη και την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών, αλλά και την ενδοοικογενειακή βία. Το Λουξεμβούργο θα επιταχύνει τι σχετικέ εργασίε προκειμένου να κυρωθεί η σύμβαση αυτή μετά την Προεδρία και ε, μια διπουργική ομάδα εργασία ήδη ασχολείται με το θέμα αυτό. Θέλουμε στο δυνατόν συντομότερα να είμαστε μεταξύ των κρατών του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν κυρώσει τη σύμβαση αυτή το Μάρτιο του 2015. Το Υπουργείο Ισότητας των Ευκαιριών υπέβαλε την πρώτη μεγάλη μελέτη που πραγματοποίησε το Luxembourg Institute of Health για τις ε, αιτίες της ενδοκογενειακή Βία στο Λουξεμβούργο. Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε μέσα σε μια διετία εντοπίζοντας ε, στοιχεία για τα θύματα, τους ε, αυτούργους και τους επαγγελματίες του χώρου. Ε, τα πορίσματα παρουσιάστηκαν στην Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας τον περασμένο Μάρτιο, στα πλαίσια μιας μεγάλης διεθνούς διάσκεψης, με συμμετοχή εθνικών και διεθνών εμπειρογνωμόνων, μελέτη που επιβεβαίωσε τη διαπίστωση ότι οι γυναίκες κατά πλειοψηφία είναι θύματα, ενώ οι άντρες ως επιτοπλίστων οι υπεύθυνοι, οι δράστες της ενδοοικογενειακής βίας. Η μελέτη δείχνει ότι ένα μία μελιτέο ποσοστό ανδρών μπορεί και αυτοί να είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ενώ αντιστοίχως ε, κάποιες γυναίκες μπορεί και αυτές να είναι δράστριες σε περιπτώσεις ε, ενδοοικογενειακής βίας. Πρόκειται για θέμα ε, πνευματικής εντιμότητας των να καταγράψουμε αυτά στις διαπιστώσεις και να συγκεντρώνουμε ε, στοιχεία προκειμένου να την αναχαιτήσουμε ε, στο δίνεκες. Ε, πιστεύουμε ότι ψυχολογική και κοινωνική πλαισίωση δεν πρέπει να απευθύνεται μόνο στα θύματα της βίας, αλλά και στους δράστες στους δράστες για να αποφύγουμε την, ε, τον υποτροπιασμό τους. Η ενδογενειακή βία είναι ένα παραλαμβανόμενο φαινόμενο στις οικογένειες. Γι' αυτό συστήνουμε στο πλαίσιο αυτό οι διεθνείς οργανώσεις ε, και τα κείμενα που εγκρίνονται από αυτές να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τις διαστάσεις αυτές, τις πτυχές αυτές που αποτελούν μέρος μιας πραγματικότητας που είναι ήδη πολύ ζωφερή και πολύ περίπλοκη. Επιπλέον διαπιστώνουμε ότι ο ορισμός της βίας εις βάρος των γυναικών, ιδίω ε, της συνδικοκαινιακής βίας, ε, διαφέρει, διαφέρει ανάλογα με το ποια διεθνής οργάνωση τον διατυπώνει. Οι ορισμοί που έχουν ε, χρησιμοποιηθεί στην Εθνική Νομοθεσία επίσης διαφέρουν. Το φαινόμενο της βίας απαιτεί διαφοροποιημένες προσεγγίσεις. Πάντως πιστεύω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για του όρου που χρησιμοποιούμε, να είναι κοινοί και οι δείκτε να είναι συγκρίσιμοι και μετρήσιμοι. Η Λουξεμβουργιανή Προεδρία χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό το σχέδιο μελέτης του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το κόστος των μορφών βίας εις βάρος των γυναικών και τις ψυχολογικές και σωματικές φθορές που μπορεί να προκαλέσουν. Βεβαίως, δεν μιλάμε μόνο για ιατρικό και νοσοκομιακό κόστος, αλλά και δικαστικό ή κοινωνικό κόστος. Ένα άλλο θέμα που σχετίζεται άμεσα με τη βία και την δεσποτεία είναι το σύνταγμα ακόμα και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητό στο πρόγραμμα της Λουξεμβουριανής Προεδρίας, διαπιστώνουμε ότι κάποια κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Γαλλία, η Γερμανία ή και κατοχώρε ε, συζητούν αυτή τη στιγμή στα κοινοβούλια τους το θέμα αυτό. Η όλη συζήτηση αφορά όλος ιδιαιτέρως ε, το να ξέρουμε ποιο είναι το νομικό πρότυπο για να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της πορνεία στην επικρατειά μας τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης συζήτησαν το θέμα και ενέκριναν ένα σχετικό ψήφισμα για την πορνεία, την εμπορία και τη σύγχρονη δουλεία στην Ευρώπη. Τοποθετήθηκαν υπέρ του σουηδικού μοντέλου που προβλέπει μεταξύ άλλων την ποινικοποίηση των ε, ε στοιχείων αυτών. Η πορνεία είναι και αυτή ένα περίπλοκο φαινόμενο που πρέπει να το συζητήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί αφορά όλα τα κρατημέλη. και τα διμερείς μας επαφές με τους συναδέλφους ε, από τις άλλες χώρες, ε, το θέμα αυτό το συζητούμε διαρκώς. Ε, το θέμα της πορνείας και της εμπορίας των ανθρώπων και ταχθήκαμε υπέρ της ενισχυμένης ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα αυτό. Κυρίες και κύριοι, ένα τελευταίο θέμα, ένα τελευταίο θέμα που δεν θα το καλύψει η Λουξεμβουργιανή Προεδρία Κάτι που μου είναι ιδιαίτερα προσφυλέ είναι αυτό των μισθολογικών αποκλήσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Οι μισθολογικέ αυτέ διαφορέ εξακολουθούν να αποτελούν πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάσει μια μελέτη τη Eurostat που δημοσιεύθηκε το Μάρτιο φέτο, ε, η απόκληση των μισθών ανδρών και γυναικών φτάνει το 16,4% κατά μέσο όρο το 2013 και 17,3% το 2008 έχει μειωθεί στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά έχει διονγκωθεί σε ε, μια δεκαριά άλλες. Οι αριθμοί τι μας δείχνουν, ότι οι στόχοι που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την προώθηση της απασχόλησης των γυναικών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Ευρώπη 2020 για να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης από 75% στο 75% στο 2020 μπορεί να συνεισφέρουν στην κάλυψη της μυθολογικής απόκλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών. Θα πρέπει ωστόσο να εντείνουμε τις προσπάθειές μας προκειμένου να εκριζώσουμε τα στερεότυπα τα οποία ε, σχετίζονται με το φύλλο, ιδίω τον επαγγελματικό βίο, για να φτάσουμε μεταξύ άλλων σε καλύτερη διαφοροποίηση των επιλογών που προσφέρονται στις γυναίκε για επαγγελματική σταδιοδρομία. Εν τέλει, είμαι πεπισμένη ότι η προώθηση των γυναικών στη διαδικασία λήψη οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων θα έχει και τι θετικέ της επιπτώσει ω προ την καταπολέμηση τη μυθολογική απόκληση ανδρών και γυναικών, η ε, ενισχυμένη παρουσία των γυναικών στου φορεί που λαμβάνουν αποφάσει μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή νοοτροπία. Μπορεί πραγματικά έτσι να φτάσουμε το στόχο μα ω προς την εργασία, ίση θέση εργασίας και ίση μισθή. Ε, σίγουρα μακρηγόρησα λίγο κυρίες και κύριοι, να με συγχωρείτε, αλλά ήθελα πραγματικά να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Λεξουμπουριανής Προεδρίας. Είμαι υπερήφανη που είμαι μαζί σας σήμερα με τη συνάδελφό μου υπουργό για, την οικογένεια, για τα οικογενειακά ζητήματα και την ένταξη και σας ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας. Είμαστε διάθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Μας παρουσιάσατε με πολλές λεπτομέρειες το πρόγραμμά σας και θίξατε τα περισσότερα ζητήματα τα οποία απασχολούν την Επιτροπή μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για την ε, μακρά παρέμβασή σας. Η κυρία Κορίν Καέν έχει τώρα το λόγο που είναι Υπουργός Οικογενειακών Υποθέσεων και Ένταξης. Και μετά θα ακούσουμε τις παρεμβάσει των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Κύριε Καέν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε και κύριοι Αντιπρόεδροι και εσείς Ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ που με προσκαλείτε να λάβω το λόγο ενώπιόν σας. Επιθυμώ να αναφερθώ στις πολιτικές εντάξεις των Ρωμά και την αντιμετώπιση του αντιαθηγανισμού. Για τις πολιτικές της Προεδρίας του Λουξεμβούργου και για το πρόγραμμά μας για την πρόθεση της ποικιλομορφίας και πολυφωνίας και του αγώνα κατά πάσης μορφής διακρίσεων. Τα τρία θεσμικά όργανα, επίσης το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι χώρες μέλη και η κοινωνία των πολιτών, όλοι έχουμε αναλάβει δέσμευση άνευ προηγουμένου για την ένταξη των Ρωμά στις κοινωνίες μας. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε λίγα παραδείγματα. Πρόσφατα, 15 Τετάρτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που ζητεί από τις χώρες μέλη να αναγνωρίσουν επισήμως τη γενοκτονία κατά των Ρωμαίων στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να ε, φτιάξουν και επέτειο, ετήσια επέτειο για το ολοκαύτωμα των Ρωμά. Αυτό έχει σημαντικό συμβολισμό και υπενθυμίζει το βαρύτατο τίμημα που κατέβαλε η κοινωνία των Ρωμά, η κοινότητα των Ρωμά, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Επίση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε την πρώτη Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Αυτά για να διευκολυνθεί μια ανταλλαγή θετικών πρακτικών και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των χωρών μέλων. Είχα την μεγάλη χαρά να συμμετάσχω στην τελευταία συνεδρίαση στις 16 Τρίτου εδώ στις Βρυξέλλες της πλατφόρμας αυτής. Επίσης το έκτακτο συμβούλιο της 19ου ε, της 19ης μάλλον συζητήθηκαν παρόμοια θέματα. Το Συμβούλιο έχει καλέσει τις χώρες μέλη να λάβουν ειδικά μέτρα υπέρ των Ρωμά σε τομείς όπως η παιδεία, εκπαίδευση, η απασχόληση, η πρόσβαση σε φροντίδες υγείας και σε στέγη και να βελτιωθεί η ε, επικοινωνία μεταξύ των κοινοτήτων Ρωμά και των τοπικών κοινωνιών. Στη βάση της συνταγματικής επιταγής ισότητας που λέει ότι όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται σε υπό τις ίδιες συνθήκες θα αντιμετωπίζονται με ισότητα. Εμείς υποστηρίζουμε την ισότιμη μεταχείριση όλων των πολιτών ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής ή εθνικότητας. Επίσης, στο Λουξεμβούργο έχουμε ανθρώπους από 160 εθνικότητες και είναι περίπου το 46% του πληθυσμού μας. 46% του πληθυσμού μας που δεν είναι Λουξεμβούργοι. Να λοιπόν γιατί ασκούμε αυτή την πολιτική. Έχουμε την ευκαιρία λοιπόν να ζήσουμε μέσα σε ένα πραγματικό χωνευτήρι εθνικοτήτων στο Λουξεμβούργο και πολιτισμών που διαχέουν ολόκληρη την λουξεμβουργική κοινωνία. Στη χώρα μου, στο Λουξεμβούργο, η ένταξη των Ρωμά αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος μιας Γενικότερη πολιτική η οποία λαμβάνει υπόψη όλες, ε, όλα τα ίδια κρίσεων βεβαίω. Το, σε 9 ε, Σεπτεμβρίου 2013 λάβαμε μέτρα για την Για, ναι, αυτά. Λοιπόν, για να ευξήσουμε τη συνεργασία, την ε, εθνική συνεργασία στον τομέα αυτό. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση των παιδιών και των γυναικών. Επίσης, το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έφεξε ένα δίκτυο σημείων επαφών για την ένταξη των Ρωμά. Οι πολιτικές υπέρ των πληθυσμών Ρωμά βρίσκουν απήχηση και στην στρατηγική της Ευρώπης για τους στόχους του 2020. Έτσι λοιπόν μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ορισμένες χώρες μέλη έλαβαν συστάσεις, δέχτηκαν συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ένταξη των Ρωμά στις κοινωνίες τους. Υπάρχει και το Συμβούλιο των Ρωμά, το οποίο δραστηριοποιείται κατά των διακρίσεων. Το, η Επιτροπή ΚΑΡΟΜ, Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, προωθεί συστάσεις για εθνικά θέματα, για εθνικά μέτρα μάλλον και για ανταλλαγή θετικών πρακτικών. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, παρόλε αυτέ τι πρωτοβουλίε, υπερβολικά μεγάλο αριθμό Ρωμά υφίσταται διακρίσει, κοινωνικό αποκλεισμό και ακόμα χειρότερα ε, εκδηλώσει μίσου. Λοιπόν, όλε αυτέ οι πολιτικέ είναι ουσιώδει. Είναι όμω επαρκή. Δυστυχώ. Η απάντηση οφείλει να είναι αρνητική. Η κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε σε ορισμένε χώρε μέλη αποδείχνει ότι έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε και ότι βρισκόμαστε ακόμα πολύ μακριά από μια κατάσταση όπου η, τα πρόσωπα ε, καταγωγή Ρωμά θα ενταχθούν πραγματικά στι κοινωνίες μα. Συμφωνώ με τη διεκδίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ληφθούν μέτρα ώστε όλα τα παιδιά, μεταξύ αυτών και τα παιδιά Ρωμά, να έχουν τα ίδια δικαιώματα, δηλαδή πρόσβαση στην εκπαίδευση, πρόσβαση σε φροντίδε υγεία σε στέγη, με λίγα λόγια σε αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης που να τους επιτρέψουν να βάλουν μια στέρεα βάση για την ενήλικη ζωή τους. Είναι επίσης σημαντικό να προωθηθούν και τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα ανδρών και γυναικών και μέσα στις κοινότητες ΡΟΜ. Δυστυχώς δεν στέφονται από επιτυχία όλες αυτές οι προσπάθειες, δεν θα στεφτούν από επιτυχία εφόσον δεν ευαισθητοποιήσουμε τις κοινωνίες να δεχθούν τις κοινότητες Ρώμ στους κόλπους τους με αξιοπρέπεια. Η ένταξη ε, βεβαίω είναι αμφίδρομη υπόθεση. Δεν αρκεί να δημιουργηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες για την ένταξη, να δημιουργηθούν τα απαραίτητα εργαλεία. Χρειάζεται και η ίδια η κοινωνία υποδοχής να κάνει μια προσπάθεια απέναντι στους ανθρώπους που επιθυμούν να ενταχθούν. Για να μπορέσουμε λοιπόν να δεχθούμε τον άλλον πρέπει να τον γνωρίζουμε και να τον καταλαβαίνουμε. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, είναι πρωταρχική σημασίας να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες απέναντι στις πραγματικότητες, στον τρόπο ζωής, στον πολιτισμό των ε, κοινοτήτων Ρωμά. Είτε έχουν εγκατασταθεί κάπου μόνιμα είτε όχι. Πρέπει να αλλάξουν οι νοοτροπίες. Πρέπει να μάθουμε να ρίχνουμε μια ματιά στον άλλο χωρίς προκαταλήψεις. Εμείς στη χώρα μου δηλαδή, πλησιάζουμε στο να φτάσουμε να δίνουμε σε όλους τα ίσα δικαιώματα ανεξαρτήτως είτε ε, καταγωγής, είτε ε, κοινωνικών, θρησκευτικών ή άλλων πεπιθήσεων, είτε ε, ερωτικής ή γενετήσιας ε, προσέγγισης κ.ο.κ. Χρειάζεται λοιπόν μια προσέγγιση συνολική. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε μονάχα σε μέτρα κοινωνική πολιτική Πρέπει να απευθυνθούμε στο πνεύμα της κοινωνίας. Κοιτά, έχω να σας εξηγήσω και δύο πρωτοβουλίες. 27 και 28 δεκάτου 2015 θα συνέλθει στο Λουξεμβούργο η High Level Group on Discrimination καθώς και το Διεθνές Φόρουμ της ε, Ισότητας. Και εκεί θα συζητηθούν θέματα διακρίσεων ισότητας μεταχειρήσεως και ευκαιριών. Στις 28 Δεκάτου θα δώσουμε ιδιαίτερο ρόλο, στο, ιδιαίτερο, ιδιαίτερη σημασία μάλλον, στον ρόλο του τύπου, καθώς επίσης και των μέσων ενημερώσεως και στον ρόλο που μπορούν να παίξουν για να αυξηθεί η αποδοχή απέναντι στις κοινότητες Ρωμά. Ο τύπος έχει σημαντικό ρόλο να παίξει και είμαι βεβαία ότι θα συζητήσουμε τα πάντα σχετικά στις 28 Δεκάτου. Είμαι πεπισμένη επίσης ότι η πολυφωνία είναι πραγματική, πραγματικός πλούτος για τις κοινωνίες μας. Πρέπει να μάθουμε να την αναγνωρίζουμε και να την αποδεχόμαστε αμοιβαία. Να γνωρίζει κανείς κάποιον άλλον σημαίνει να μπορεί να κατανοεί και το παρελθόν του και την ιστορία του. Το ψήφισμα που ενέκρινε στις 15 Τετάρτου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς εκεί κατευθύνεται. Επίσης το Συμβούλιο Υπουργών έχει ταχθεί κατ' επανάληψη κατά των διακρίσεων σε βάρος των Ρωμά δεν έχει τοποθετηθεί σχετικά με την ε, ετήσια επέτειο της γενοκτωσίας του ονομά. Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι η καλύτερη κατανόηση της ιστορίας ε, βοηθεί, συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση. Επίσης, η μελέτη του παρελθόντος θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το παρόν. Η ιστορία των Ρωμά συναποτελεί μέρος της δικής μας ιστορίας. Ο πολιτισμός των Ρωμά πρέπει να γίνει μέρος του δικού μας πολιτισμού. Πρέπει να μπορέσουν να ενταχθούν στις κοινωνίες μας διαρκής διάλογος μεταξύ των διαφόρων θεσμικών μας οργάνων, συντονισμός, ενισχυμένος συντονισμός, θα ωφελήσει τις πολιτικές των χωρών μελών, καθώς επίσης και τις κοινότητες Ρώμα. Είμαι απόλυτα πεπισμένη περί αυτού. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτέ, είμαι πραγματικά πολύ ικανοποιημένη που βρίσκομαι ενώπιον σας σήμερα και σας ευχαριστώ ιδιαίτερως για την προσοχή σας. Είμαι βεβαίως στη διάθεσή σας εφόσον επιθυμείτε να θέσετε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και τις δύο υπουργούς για τις παρουσιάσεις τους που ήταν τόσο πλήρης όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες. Περνάμε λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις και απαντήσεις. Έχουμε δέκα συναδέρφους στον κατάλογο μιλητών μέχρι τώρα. Αρχίζουμε με τους πρώτους πέντε, μετά θα πάρουν το λόγο οι υπουργοί και μετά οι υπόλοιποι. Κόστιγκερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ και τις υπουργούς για την εκτεταμένη περιγραφή του προγραμματός νομίζω ότι πολλά από όσα είπαν έπεσαν σε γόνιμο έδαφος, ομιλώ και εξ ονόματος της συντονίστριάς μας Λεγκρίπ. Για εμάς, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, πολύ σημαντικές είναι οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό. Ήδη μιλήσατε σχετικά. Ο ρυθμός απασχόλησης των γυναικών πρέπει να επεκταθεί και βεβαίως θα καταβάλουμε και άλλες προσπάθειες από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κάνουμε ό,τι μπορούμε. Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να είναι ένα πρόβλημα. Όπως είπατε υπάρχει ανάγκη να θεσπιστούν ίσες αμοιβέ για ίση εργασία. Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών μελών. Όμως ο μέσος όρος φτάνει το 60% της αμοιβή της γυναικός έναντι της αμοιβή του ανδρός. Ακόμα μεγαλύτερο είναι, το, είναι η απόσταση στις συντάξεις Ο μέσο όρο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι τη τάξη του 38%. Η ε, κυρία Ζαμπόρσκα κάνει και μια σχετική έκθεση και έχει εξετάσει το θέμα και ελπίζουμε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με το ε, Συμβούλιο Υπουργών έτσι ώστε να προωθήσουμε μια ρύθμιση για τον εξυγχρονισμό και το κλείσιμο των κενών. Στο πρόγραμμά σας αναφέρεστε και στην ανάγκη ισότιμης εκπροσώπησης και στα διάφορα πολιτικά όργανα και επίσης όργανα λήψης αποφάσεων. Εδώ θέτω ερώτηση. Τι γίνεται με την οδηγία Women on Boards του Συμβουλίου. Έχουμε κάνει προτάσεις σε μια πρώτη ανάγνωση. Το αποτέλεσμα υποστηρίζεται από τις μεγάλες ε, κοινοβουλευτικές ομάδες. Τι προτίθεστε να πράξετε για να οδηγήσετε σε μια αίσια έκβαση την ε, οδηγία αυτή. Επίσης, πρόσφατα μιλήσατε μάλλον και για την κύρωση της ε, συνθήκης της Ισταμπούλ. Και εδώ με ενδιαφέρει να μάθω ποιες είναι οι προσδοκίες σας. Τι θα πράξει η Λουξεμβουργική Προεδρία πιο συγκεκριμένα για να επιτύχει τον στόχο αυτό. Και εδώ όλες νομίζω συμφωνούμε ότι είναι σημαντικό να γίνουν ορισμένες προσπάθειε. Ορισμένε ε, χώρε μέλη έχουν ήδη υπογράψει και λένε ότι η βία κατά των γυναικών, ο αγώνας δηλαδή κατά της βίας κατά των γυναικών πρέπει να είναι υψίστη προτεραιότητα. Και εδώ θα ήθελα να ακούσω πιο συγκεκριμένα πράγματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εσεί τώρα κυρία Χόνιμπολ. Ευχαριστώ. Εκ μέρου τη Μαρία Σαρένα που είναι συντονίστριά μας αλλά δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πολύ για την τόσο πλήρη παρουσίαση της καθεμιάς σας για το τι κάνετε. Πραγματικά σας ακούσαμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση και βλέπουμε ότι η Προεδρία σας παίρνει πολύ σοβαρά το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών. Θα σας ε, διαβάσω αυτά που έχω από την κυρία Ρένα πρώτα απ' όλα που έχουν ως Στις προτεραιότητές σας αναφέρεται ότι θα δώσετε ιδιαίτερη σημασία στην απασχόληση των γυναικών. Αν θέλετε να την ενισχύσετε πρέπει να πάρετε μέτρα για να ε, μπορέσουν οι γυναίκες να συνδυάσουν καλύτερα την επαγγελματική με την προσωπική του ζωή. Πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ε, άδειας μετά τον τοκετό. Το θέμα αυτό ξέρουμε πόσο πολύ έχει δυσκολέψει τους ευρωβουλευτές και ξέρουμε πόσες προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι τώρα για να αρχίσει και πάλι ο διάλογος μετά τις μέχρι τώρα αποτυχίες. Πράγματι είναι ένα θέμα που πειράζει πάρα πολύ την ε, ισορροπία στα δικαιώματα ανδρών και γυναικών. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν σχετική νομοθέτηση. Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών δεν έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα. Τώρα βιαζόμαστε, πρέπει να ενισχυθεί η απασχόληση των γυναικών και η γονιμότητα επίσης. Θέλουμε λοιπόν προτάσεις μέχρι τα τέλη του μήνα, όμως δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες. Θέλουμε λοιπόν να ξέρουμε εσείς πως έχετε περισσότερες πληροφορίες για το τι κάνει η Κομισιόν από αυτού και τι θα κάνετε για να στηρίξετε φιλόδοξα νομοθετικά μέτρα προκειμένου να συνδυαστεί καλύτερα η ζωή των γυναικών στο επαγγελματικό και το προσωπικό επίπεδο και τι θα κάνετε για τη μητρική άδεια. Επιτρέψτε μου επίσης να προσθέσω και κάτι ένα δικό μου σχόλιο που έχει να κάνει με την πορνεία και την ε, εκμετάλλευση των γυναικών. Την λαθροδιακίνηση. Ξέρετε ότι έχουμε κάποιο συντονιστή από αυτού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη Δευτέρα που μας πέρασε ενέκρινε έκθεση όσον αφορά το θέμα της πορνείας ακριβώς, όπου συστήνουμε να ακολουθήσουμε το σουδικό μοντέλο. Οπότε χαίρομαι πολύ που η δικιά σας Προεδρία ασχολείται με αυτό το θέμα. Σας ανθαρρύνω να συνεχίσετε να το κάνετε, γιατί δεν μπορούμε να πετύχουμε συμφωνία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά τα τόσο δύσκολα και περίπλοκα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πορνεία και την λαθρέα διακίνηση ατόμων. Η κυρία Ζνιάσκα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πραγματικά Πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πολύ που σας έχουμε εδώ μαζί μας. Σας ακούσαμε. Χαιρόμαστε που έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας. Σας ακούσαμε για τα διάφορα ζητήματα, διαφορές στους μισθούς μεταξύ ανδρών και γυναικών και άλλα. Ε, να ξέρετε ότι εκτιμώ όλους ιδιαίτερο την παρέμβαση της κυρίας Καέν που αναφέρθηκε στο ζήτημα των διακρίσεων αυτών. Με εξέπληξε, ήταν κάτι που δεν είχα βρει στις προτεραιότητές σας, οπότε πολύ χάρηκα που σας άκουσα. Γιατί είναι ένα θέμα που στη χώρα μου είναι πολύ σημαντικό, βλέπετε, και πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης συζητιέται ήδη, αλλά δυστυχώς χωρίς να καταλήγουμε σε λύση. Πρέπει να βρούμε λοιπόν συγκεκριμένα εργαλεία για να καταλήξουμε και σε λύση. Έρχομαι τώρα στις ερωτήσεις μου. Ίσες ευκαιρίες. Αναφερθήκατε στην κοινωνική διάσταση και λέτε ότι θέλετε να επικεντρωθείτε κυρίως στα άτομα εκείνα τα οποία είναι πιο ευάλωτα που χρειάζονται περίθαλψη ή οτιδήποτε άλλο. Θέλω να γνωρίζω λοιπόν ποιο είναι το σημείο κίνησης που έχει η δικιά σας Προεδρία για αυτό το ζήτημα. Γιατί είναι σημαντικό στα πλαίσια της βελτίωσης της περίθαλψης των ατόμων εκείνων, για παράδειγμα, που ζητιανεύουν. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο ζήτημα, στο θέμα της παιδείας. Εδώ θέλουμε δομές για την, για, την, για, την, για τα μικρά παιδιά. Θέλουμε θεσμούς ποιότητας που να ασχολούνται με τα παιδιά. Υπεύθυνα για την παιδική μέρημνα. Έπειτα, Κάτι άλλο, πώς θα διασφαλίσουμε πραγματική πρόσβαση στην δικαιοσύνη για τα παιδιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ συγκεκριμένες οι ερωτήσεις αυτές. Έχουμε μισή ώρα ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί η συνεδρίασή μας. Οπότε να συμφωνήσουμε το εξή. Θα δώσουμε το λόγο σε όσους έχουν ερωτήσεις και μετά θα δώσουμε το λόγο στις υπουργού για να απαντήσουν. Ελπίζω έτσι να μπορέσουμε να τα προλάβουμε όλα μέσα στη μισή ώρα που μας μένει. Παρακαλώ, επόμενη ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη και ευχαριστώ τις υπουργούς που ήρθαν να μας μιλήσουν σήμερα για τις προτεραιότητες της Λουξεμβουργιανής Προεδρίας. Νομίζω ότι όλοι χαρήκαμε να ακούσουμε πόσα πολλά έχετε σκοπό να κάνετε, διότι οι δύο-τρεις γραμμές του προγραμματός σας ήδη απηχούν την διάθεσή σας ως προς τα ζητήματα των γυναικών, είναι λοιπόν καλύτερο να μπορούμε να ακούσουμε μια εκτεταμένη εκδοχή των όσων έχετε σκοπό να κάνετε. Και τον Δεκέμβριο θα περιμένουμε ανυπόμονα να δούμε πόσο θα έχετε επιτύχει. Χάρηκα ιδιαίτερα που άκουσα ότι θα επικεντρωθείτε και στις ευρωεκλογέ και την επιλογή των υποψηφίων αλλά και για τους Ρωμά ένα θέμα που και αυτό με απασχόλησε και επειδή το θέμα με τους Ρωμά έχει να κάνει και με την διακίνηση και εμπορία. Η πλειοψηφία των παιδιών που διακινούνται ανά την Ευρώπη είναι παιδιά των Ρωμά και είναι αποτέλεσμα της φτώχειας. Πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσει η εμπορία παιδιών. Το 2013 το Κοινοβούλιο υιοθέτησε την ε, ατζέντα του για την ισορροπή εκπροσώπηση των γυναικών της εταιρεία που είναι συγμένες στο χρηματιστήριο. Και ε, δυστυχώς αυτό δεν προχώρησε όσο θέλαμε. Απογοητευτήκαμε πολύ γιατί δεν έχει υλοποιηθεί η σχετική μας σύσταση και γνωμοδότηση για την θέση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια Θα το γνωρίζετε λοιπόν αυτό παρά τι απελπισμένε μα προσπάθειε, τι απέλπιδε προσπάθειε τη Επιτροπή μα να προχωρήσει αυτό το θέμα. Τελικά δεν έχει προχωρήσει αρκετά. Οι γυναίκε στα διοικητικά συμβούλια λοιπόν, αυτή η πρόταση μπορεί να επανέλθει. Θα μπορούσε να εξεταστεί με μεγαλύτερη προσοχή για το Συμβούλιο. Θα σα είμαστε ευγνώμονε και θα σταματήσω εδώ. Έχω κι άλλα να πω, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν κι άλλοι που θέλουν να πάρουν τον λόγο. Ευχαριστούμε κυρία Μπιόρκ. Ευχαριστώ και τις δύο υπουργούς για το φιλόδοξο πρόγραμμα και τα σχόλια που έκαναν. Η Προεδρία του Λουξεμβούργου φέρνει την οικογένεια και τα ζητήματα, τις υποθέσεις της οικογένειας μεταξύ των προτεραιοτήτων της. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε μία από όλες αυτές τις πτυχές. Η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών είναι κάτι που το αναφέρατε και οι ίδιες. Μπορεί οι πολιτικές λιτότητας εδώ να έχουν κάποιον αντίκτυπο και η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών να πλήττεται από αυτές. Αυτό πιστεύω πρέπει να συζητηθεί πιο έντονα στο επίπεδο του Συμβουλίου και χρειαζόμαστε δείκτες για το πώς έχει μεταβληθεί η κατάσταση στις χώρες που έχουν εκτεθεί στις πιο αυστηρές πολιτικές λιτότητας. Ως προς τους στόχους μας για τα παιδιά. Δεν είδα καμιά ιδιαίτερα φιλόδοξη προσπάθεια για να προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε τη σχετική περίφερψη. Αυτό είναι σημαντικό για την ισότητα, αλλά και για τους άνδρες και την ισότητα. Το φθινόπωρο θα οργανωθεί ένα σχετικό εργαστήριο άνδρες και ισότητα. Και προοπτική των φεμινιστριών προ αυτό. Φυσικά και υπάρχει διακριτική μεταχείριση των ανδρών σε κάποιε χώρε. Οι άντρε δεν έχουν δικαίωμα σε γονική άδεια, δε, λόγου χάρη. ή ο τρόπο που τα στερεότυπα και για τους άντρε δομούνται, ε, η δράση των ανδρών για την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών είναι όλα στοιχεία που πρέπει να τα δούμε με μεγαλύτερη προσοχή. Πώ μπορούν οι άντρε να προλάβουν τη βία κατά των γυναικών. Εν τέλει, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια για τι γυναίκε και την ισότητα στι εξωτερικέ μα πολιτικέ, Στι εξωτερικέ μα δράσει. Αν δείτε τα κονδύλια που προβλέπονται για τα όσα πρέπει να γίνουν για την ισότητα και την ισότητα των γυναικών κυρίω, τα κονδύλια αυτά είναι μηδαμινά. Εγκρίναμε την έκθεση Νόχλη για τη θετική τη ισότητα σχετικά πρόσφατα και υπήρχαν εκεί πολύ καλέ συστάσει που καλό θα ήταν να ακολουθηθούν. Νομίζω όμως ότι είναι σημαντικό όλοι οι Υπουργοί Ισότητας, εφόσον υπάρχουν αρμόδιοι Υπουργοί, να συναντηθούν και να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα στο Συμβούλιο για την προώθηση και την προβολή των θεμάτων αυτών. Υπουργέ θα είμαστε κοντά σα για να αντιμετωπίσουμε τα φαινόμενα αντιαθηγανισμού και την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάποιοι θεωρούν ότι αρκεί η ανεκτικότητα. Όχι, χρειάζεται δικαιοσύνη και ισότητα. Αυτό σημαίνει και στέγαση και πρόσβαση στην εκπαίδευση και θέσει εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Μπιόρκ. Ο λόγο στην κυρία Ράινστρο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μούτς, κυρία Καν. Εκ μέρου των Πρεσίνων παίρνω το λόγο σήμερα. Δουλεύουμε για τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. COP21. Δεν θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τις προκλήσεις που έχουν να κάνουν με το κλίμα αν δεν επικεντρωθούμε και στο ζήτημα της ισότητας των φύλων. Έχετε αναφερθεί πολύ στη διάσταση του φίλου σε όλες τις πολιτικές μας. Η ερώτηση μου λοιπόν έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή ακριβώς. Και με αυτή τη συνάντηση στο Παρίσι. Η Λουξεμβουργιανή Προεδρία. Τι πολιτική έχει και τι στρατηγική έχει για την περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Κυρίως όσον αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας σε αυτές τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία για το Κλίμα. Ξέρουμε ότι ο λόγος για τη διάσταση του φύλου και την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων είναι κάτι πολύ σημαντικό και είναι βασικό έτσι ώστε τα μέτρα χρηματοδότησης για την προσαρμογή εξαιτίας της αλλαγής του κλίματος πρέπει να φροντίσει και τους πιο φτωχούς και τις γυναίκες, κυρίως στο Νότο. Η κυρία Ρόμπινσον δουλεύει πάνω σε αυτό το θέμα για την εκπροσώπηση των γυναικών και για πολιτικές που είναι ευαίσθητες στο θέμα της διάστασης του φύλου. Συνεπώς, ρωτάω, θα είναι προτεραιότητά σας να μιλήσετε για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των δύο φίλων στην τελική συμφωνία που θα επιτευχθεί στο Παρίσι. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Γιούτεχ, τώρα το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ ιδιαίτερα στους υπουργού για τις ομιλίες τους διότι πραγματικά αισθανθήκαμε και εμείς τον ενθουσιασμό σας ε, για τα θέματα που καλύψατε. Εγώ μιλώ εξ ονόματος της ομάδας CFTD e και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη για να μπορέσετε να απαντήσετε. Ναι, όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο. Ένα μεγάλο θέμα που δεν νομίζω ότι το αναφέρατε, ίσως λόγω έλλειψης χρόνου, είναι το αν θα υπάρξει κάποια πολιτική ενέργεια, κάποιο πρόγραμμα, κάποια πρόθεση που μπορεί να έχει η Προεδρία σας για να ασχοληθεί με τις μορφές βίας και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τρίτες, των γυναικών από τρίτες χώρες. Μεταξύ των προθέσεων της Προεδρίας σας κάποια δράση, κάποιο μορφή προστασία, κάτι σκοπεύετε να οργανώσετε για τις συγκεκριμένε αυτές μορφές βίας στα βασανιστήρια, αλλά μιλώ χάρη για, τις, ε, για τους λιθοβολισμούς κατά των γυναικών και περιπτώσεις που πολύ συχνά αποσιωπούνται. Αυτό είναι η πρώτη μου ερώτηση, αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση και έπειτα το επενήχθησαν και άλλες συνάδελφοι σε σχέση με την οδηγία για την άδεια μητρότητας. Φεύγουμε από ένα εξάμεινο όπου η Προεδρία μας απογοήτευσε Ελπίζω η στάση σας να είναι στάση μεγαλύτερης συνεργασίας ε, με την Επιτροπή μας, πιο θετική. Και πραγματικά ελπίζω να δώσουμε σάρκα και οστά σε, αυτό το, σε αυτή την πρόθεση που αναφέρατε. Λείπει η οδηγία αυτή, χρειάζεται να γίνει μια νέα αρχή, αλλά ερώτηση είναι αν έχετε ήδη επιταπτώσει κάτι συγκεκριμένο, εάν σε αυτήν την νέα αρχή έχετε ήδη δώσει μια έκφραση. Διότι οι μαμάδες σε όλη την Ευρώπη περιμένουν απελπισμένα την έκβαση της πορείας αυτής της οδηγίας. Ευχαριστούμε η κυρία Μίλναρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τις κυρίες Υπουργούς. Συγκεκριμένη ερώτηση. Συνθήκη της Ισταμπούλ που είναι το πρώτο νομικά δεσμευτικό έγγραφο για την καταπολέμηση πάσης μορφής βίας κατά γυναικών και ε, νέων κοριτσιών εγκρίθηκαν εγκρίθηκε μάλλον από τα 47 κράτη-μέλη και άρχισε να ισχύει από το 2014. Μέχρι τώρα όμως μόνο 9 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχουν κυρώσει. Μάλιστα ορισμένες χώρες μέλη κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Για παράδειγμα η Ουγγαρία που έχει αποκλείσει το θέμα αυτό από την ημερήσια διάταξη του Ουγγρικού Κοινοβουλίου. Ενθαρρύνουμε όλες τις χώρες μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράψουν την συνθήκη αυτή. Αυτό η σύμβαση. Αυτό που θέλουμε να μάθουμε από εσά είναι τι προτίθεται να κάνει η Προεδρία σας και στο επίπεδο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο επίπεδο της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2, το Συμβούλιο μπορεί να εξουσιοδοτήσει την έναρξη διαπραγματεύσεων. Έχετε κάποια σχέδια και πού βρίσκεστε. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μιλνάρ. Η ε, κυρία Λινκεβιτσιούτε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Επιθυμώ να ευχαριστήσω τις δύο υπουργού για την παρουσίαση των θεμάτων της Προεδρίας τους. Συμφωνώ με την ενίσχυση της πιο ισορροπημένης συμμετοχής ανδρών και γυναικών στο επίπεδο λήψος αποφάσεων. Μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική. Επίσης αυτό με ενδιαφέρει. Ακόμα τα πράγματα αυτά βασίζονται σε βέλτιστες πρακτικές. Προβλέπετε να ασχοληθείτε και με κάτι άλλο εκτός από τις βέλτιστες πρακτικές. Τώρα, για να εξασφαλιστεί ότι μέχρι και 40% των θέσεων σε υψηλό επίπεδο του δημόσιου τομέα θα καλύπτονται από γυναίκες μέχρι το 2019. Πώς θα το εξασφαλίσετε αυτό και πώς αυτό θα συμβαδίζει με την οδηγία που έχει γίνει το Κοινοβούλιο για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Θεωρείτε ότι θα σας υποστηρίξουν όλες οι χώρες μέλη στην οδηγία αυτή. Άλλη ερώτηση. Ίση αμοιβή για ίση εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτό είναι μια ιστορία χωρίς τέλος πραγματικά και δεν το έχουμε λύσει το πρόβλημα πώς μπορούμε να επιτύχουμε την ισότητα. Μήπως χρειαζόμαστε οδηγία, διότι χωρίς οδηγία μου φαίνεται πολύ δύσκολο να διασφαλίσουμε την ισότητα αμοιβών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάρα Μπέλα. Κύριε Υπουργέ, κύριες Υπουργοί, αναφερθήκατε στη Συμφωνία της Κωνσταντινούπολης και άλλοι ρώτησαν γι' αυτό. Όμως εδώ στο Κοινοβούλιο δύο φορές και το 2010 για πρώτη φορά και το 2015 για δεύτερη φορά μια πλειοψηφία συναδέρφων εκφράστηκαν προκειμένου να αφιερώσουμε ένα έτος στην βία σε βάρος των γυναικών. Με γραπτή δήλωση. Σπάνια παίρνουν πλειοψηφία τέτοιες γραπτές δηλώσεις στο Κοινοβούλιο, συμβολικά. Θάξιζε τον κόπο, όμως, ώστε να επιστήσουμε την προσοχή του κόσμου σε αυτό το θέμα που είναι ταμπού σε κάποιες χώρες μέλη. Και επειδή δεν μπορούν όλα να είναι προτεραιότητες, το κάτω-κάτω γι' αυτό και μιλάμε για προτεραιότητες, μήπως μπορείτε να αντισταθμίσετε το γεγονός το ότι δεν βρίσκεται στις προτεραιότητές σας και το εξηγήσατε ότι είναι μια θεματική που έχει να κάνει με την καθημερινότητα, τουλάχιστον στο επίπεδό σας, έχοντας την Προεδρία αυτό το εξάμεινο, άλλους 5,5 μήνες, να μπορέσετε να επιστήσετε την προσοχή σε αυτό, ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ακόμη και αν δεν το κάνει για το 2016, ας είναι το 2017, να είναι το έτος για την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών μια που πρόκειται για ένα καταστροφικό πραγματικά φαινόμενο. Ευχαριστώ. σε ευχαριστούμε. Η κυρία Κολόνσκα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ τις δύο υπουργού. Πρώτα απ' όλα, μου αρέσει πάρα πολύ ο ενθουσιασμός με τον οποίο μας μιλήσατε και συμφωνώ με όλα όσα είπατε και οι δυο σας. Και σας ευχαριστώ πολύ που αναφέρεστε στο θέμα αυτό της ισότητας με τέτοια σοβαρότητα και ελπίζω να μεταφέρετε αυτή την ατμόσφαιρα, αυτό το κλίμα και στους υπόλοιπους υπουργούς. Δεν το περίμενα. Πάντως, το θέμα των ε, Αθήγανων είναι πολύ σημαντικό. Στην Πολωνία το 2011 αποφασίσαμε ότι η Δευτέρα Αυγούστου θα είναι μια ημέρα κατά την οποία θα τους τιμούμε, γιατί πέρασανε και αυτοί από το Auschwitz καλού. Είναι μια ημερομηνία που είναι βέβαια στις διακοπές και είναι δύσκολο να συμμετέχουν οι πολιτικοί, για παράδειγμα, σε δράσεις τέτοιες μνήμης. Όμως υπάρχει Ίσως δεν είναι η καλύτερη ημερομηνία που μπορούσαμε να διαλέξουμε, αλλά υπάρχει πάντως. Τώρα για την οδηγία. Η Επίτροπος Ρέντινγκ ε, θίγει το θέμα της επικουρικότητας εδώ. Και ίσως τελικά δεν μπορέσουμε να συνεχίσουμε, φτάσουμε σαν διέξοδο. Όμως τις χρειαζόμαστε τις ποσοστώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα θα πρέπει να σταθούν δίπλα μας για να καταπολεμηθούν αυτή οι αόρατοι φραγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι χώρες μέλη και εμείς πρέπει να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης που αναφερθήκατε στις γυναίκες που δουλεύουν και τι γίνεται όταν ε, είναι σε φάση πρόσληψης οι γυναίκες αλλά και σε φάση συνταξιοδότησης. Υπάρχουν διαφορές, γι' αυτό και πρέπει να προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Τέλος. Όσον αφορά την άδεια πατρότητας. Είναι σημαντικό. Όσο περισσότεροι άντρες παίρνουν τέτοια άδεια πατρότητας και μένουν στο σπίτι, τόσο πιο εύκολο θα είναι να είναι άντρες οι οποίοι θα μάθουν να δραστηριοποιούνται και στον οικοκυριό και στο σπίτι και έτσι οι γυναίκες να μπορούν να βρίσκονται στην αγορά εργασίας. Όλα αυτά πρέπει να τα προωθήσουμε. Σας παρακαλώ σεβαστείτε το δικαίωμα των γυναικών, τα δικαιώματα των ανδρών. Είμαστε όλοι ενωμένοι για να προχωρήσουν αυτά τα θέματα και να βρεθεί μια λύση. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα μας είπατε. Σας στηρίζω και θεωρώ ότι το πρόγραμμα εργασίας σας είναι πολύ καλό. Σαπό. Η κυρία μου το έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω τις ευχαριστίες μου αυτές των προηγουμένων για την παρουσία σας σήμερα. Δεν θέλω να επαναλάβω τα πολλαπλά σχόλια που έγιναν για την απόσταση της οδηγίας, για την αδιαμετρότητας και τις συνέπειες. Μπορούμε να κάτσουμε να συζητάμε τη θέση των γυναικών στην αγορά εργασία, το τι προβλήματα υπάρχουν ώστε οι γυναίκες να μπορέσουν να αναπτύξουν και να ε, το δυναμικό τους, αλλά αυτό θα πάρει μια δεκαετία εάν δεν αρχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράση και να πετυχαίνουμε αποτελέσματα προχωρώντας στην επιδίωξη αυτών των στόχων. Κάθε φορά που κάτι ανακύπτει θα αντιμετωπίζουμε ξανά και ξανά το πρόβλημα της οδηγίας μητρότητας που δεν θα έχει απειληθεί. Διότι έλλειψε η στήριξη για την πρόθεση της οδηγίας αυτής. Καλωσορίζω λοιπόν τα σχόλιά σας για το πώς μπορεί να πιέσετε για να ξανασυζητηθεί η οδηγία αυτή. Η δεύτερη παρατηρήσή μου έχει να κάνει με την ικανοποίησή μου για την άμεση ε, ενασχόλησή σας με το θέμα των γυναικών Ρωμά. και το τι μπορεί να γίνει γενικότερα με τις γυναίκες από εθνωτικές μειονότητες. Διότι σε όλες μας τις κοινότητες οι γυναίκες έχουν ε, διπλό πρόβλημα εφόσον προέρχονται από κάποια εθνωτική μειονότητα. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα ζητήματα βεβαίως για τον πληθυσμό των Ρωμά, όμως το ερώτημα είναι εάν θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε γενικότερα τα αποτελέσματα του έργου σας. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ρέινερ είναι η τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Λουξεμβουργική Προεδρία μόλις άρχισε. Παρ' όλα αυτά, τώρα που είμαστε ακόμα σχεδόν αρχές Ιουλίου, επιθυμώ να ευχαριστήσω την κυρία Μούτς διότι οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την Προεδρία είναι πολύ σημαντικές και εκείνο το fine-tuning σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις. Θέλω να μιλήσω τώρα για την έκθεση άνδρες και γυναίκες ισότητα φύλων στα διοικητικά συμβούλια. Ειδικά σε περίοδους κρίσεως είναι ακόμα πιο σημαντικό να τίθεται και να συζητούνται τα θέματα της πολιτικής ισότητας. Χτες το απόγευμα στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων είχαμε ως προσκεκλημένη την κυρία Γιώηροβα, η οποία μίλησε ακριβώς για αυτές τις τεχνικές λεπτομέρειες που μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για βελτιώσεις. Έτσι λοιπόν έχω ερώτηση, αλλά όχι τόσο ερώτηση, αλλά μάλλον παράκληση και πρόσκληση να συνεχίσετε να εργάζεστε επ' αυτών και ιδίως ό,τι αφορά την εργασία δημοσιότητας εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο, ήδη στην κοινοβουλευτική αυτή περίοδο που διατρέχουμε, έχουμε ψηφίσει ορισμένες εκθέσεις. Και σπρώχνουμε το θέμα αυτό, γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, αλλά και άντρες βέβαια, δεν λέω, ε, όλο και περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Ρέγνερ. Για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, η οποία ήταν σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσα και μας έδωσε την ευκαιρία να θέσουμε επιτάπητος διάφορα ζητήματα που για μας, Επιτροπή Δικαιωμάτων της Γυναίκας, έχουν μεγάλη σημασία, θα σας δώσω και πάλι το λόγο στις δύο υπουργούς, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε στη διάθεσή μας λίγο χρόνο. Αν μπορείτε, έξι λεπτά η καθεμία. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε να συναντιόμαστε στην Επιτροπή μας εδώ. Ποια θέλει να αρχίσει. Παρακαλώ, η κυρία Μούσου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρα. Έξι λεπτά είναι λίγα, αλλά θα προσπαθήσω. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις σας, πολύ ενδιαφέρουσες όλες και για τις δυο μας. Πολλοί επικεντρώθηκαν στο θέμα της οδηγίας για τις ποσοστώσεις, που είναι προτεραιότητα για τη Λουξεμβουριανή Προεδρία. Ελπίζω να πετύχουμε, να έχουμε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Όταν συζητάμε με τα συνδικάτα ή με τα επιμελητήρια στο Λουξεμβούργο μας λένε ότι αφορά λίγες γυναίκες σε απόλυτους αριθμούς. Η προβολή όμως είναι τεράστια και ο συμβολισμός είναι τεράστιος αν καταφέρουμε να προχωρήσουμε αυτή την οδηγία. Θέλω να επιβεβαιώσω το στόχο του 40%. Δεν πιστεύω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε περισσότερες υποχωρήσεις σε σχέση με το σημερινό κείμενο και το 40% που προτείνουμε. Θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε περισσότερο σε συζητήσεις για ενδεχόμενες παρεκκλήσεις, ώστε αν μια χώρα έχει ήδη βρει εθνικές λύσεις, να μην υπάρχει κίνδυνος να πληγεί η κατάσταση εκεί. Πάντως έχουμε μεγάλη στήριξη. Και θα διασφαλίσουμε οι τελευταίες χώρες οι οποίες έχουν εκφράσει επιφύλαξη εξέτασης να συμφωνήσουν τελικά μαζί μας. Αυτός είναι ο γόνος που δίνουμε γιατί μία αμφισβήτηση του ποσοστού θέτεται υπό αμφισβήτηση τη συμφωνία που έχουμε με τόσες δυσκολίες ήδη βρει με τις υπόλοιπες χώρες μέλη. Οπότε δουλεύουμε τώρα για αυτή τη ρήτρα ευελιξίας. Κατά τα άλλα θα πιέσουμε. Ελπίζουμε να έχουμε τον Οκτώβριο συμπεράσματα ή το πολύ το Δεκέμβριο σε επίσημο συμβούλιο. Τώρα για τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Πολύ αναφερθήκατε σε αυτήν. Ξέρετε ότι η επικύρωση είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών, των επιμέρους χωρών μελών. 11 χώρες μέλη έχουν ήδη πει ότι συμφωνούν το πολιτικό μήνυμα, το ισχυρό που μπορούμε εμείς να στείλουμε ως Προεδρία είναι να απευθυνθούμε στις υπόλοιπες χώρες και στο Λουξεμβούργο που δεν έχουν ακόμα επικυρώσει αλλά που θα το κάνουν εμείς μετά την Προεδρία θα το κάνουμε είναι λοιπόν μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμείς πάντως στηρίζουμε την ιδέα του να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό έτος ε, κατά της βίας σε βάρος των γυναικών, όπως πρότεινε ο κύριος Ταραμπέλα. Θέλουμε όμως το μήνυμα αυτό να το στείλουμε και να είναι ηχηρό. Όσον αφορά τώρα τη βία, και αυτό έχει να κάνει ακριβώ με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, έχουμε το πρόγραμμά μας, το τρίο, και θέλουμε να στηρίξουμε διεθνείς εκστρατείες, μεταξύ άλλων και την White Ribbon που ενθαρρύνει και τους άντρες να τοποθετηθούν σε σχέση με την προβληματική αυτή της βίας σε βάρος των γυναικών. Θα ήταν σημαντικό κάτι τέτοιο. Και μπορούμε να δεσμευτούμε σε συνεργασία μαζί σας για να πιέσουμε τόσο στα πλαίσια της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης αλλά και όσο άλλες εργασίες που γίνονται για την καταπολέμηση της βίας σε βάρος των γυναικών. Με ρωτήσατε πώς μπορούμε να αποφύγουμε να υποφέρουν περισσότερο οι γυναίκες από τις οικονομικές κρίσεις. Εδώ θα έλεγα ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε στις συζητήσεις μας κάποιες, ε, κάποιο, ένα μόνιμο έλεγχο ώστε να μπορούμε να αναλύουμε αναφύλο, δηλαδή τα στατιστικά δεδομένα που έχουμε στην οικονομία, στην απασχόληση, στην ισότητα μισθών, συντάξεις επίσης, αλλά και όσον αφορά την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, να ζητήσουμε στατιστικά δεδομένα αναφύλλω. Πρέπει δηλαδή να γίνει εδώ προσπάθεια και σε εθνικό επίπεδο, σε υπουργικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο βέβαια, ώστε να μπορούμε να ε, ανταλλάσσουμε τις βέλτιστες πρακτικές μεταξύ μας για να ενθαρρύνουμε όλους τους παράγοντες και τους φορείς να εμπλακούν υπέρ αυτής της ανάλυσης. Τώρα για το θέμα της άδειας μητρότητας. Η συνάδελφο σίγουρα θα αναφερθεί σε αυτό και για τη γονική άδεια γενικά και για το πώς συμμετέχουν οι άντρες. Εννοείται ότι ως Προεδρία καταδικάζουμε το γεγονός ότι δεν έχει συμπεριληφθεί αυτό. Ήμασταν αδύναμοι. Πριν αρχίσει η Προεδρία μας δεν μπορούσαμε να επηρεάσουμε τα πράγματα περισσότερο. Όμως επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε υπέρ και ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί σας όσο γίνεται πιο σύντομα να μας παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο. Έχουμε τακτικά επαφή με σας, με τους αρμόδιους επιτρόπους και πιστεύουμε και εμείς ότι είναι σημαντικό να αναφερθούμε στα δικαιώματα της γυναίκας και στις ευθύνες των ανδρών. Πώς θα σπάσουμε τα στερεότυπα. Ε, πολύ σημαντικό και για να συμφιλειωθεί η επαγγελματική με την προσωπική ζωή. Θα σας τα πει η συνάδελφος. Ρωτήσατε επίσης κάτι για την παραβίαση των δικαιωμάτων των αντρών. Όχι μόνο, δηλαδή, δεν αφαιρθήκατε μόνο στην διάκριση σε βάρος των γυναικών, αλλά και για θέματα όπως έχει να κάνει ο λιθοβολισμός, ο αποκεφαλισμός κτλ. Υπάρχει υπουργό για τη συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια. Εδώ πρέπει να δουλέψουμε για το Women Empowerment. Πώς δηλαδή στις χώρες αυτές θα προχωρήσει η παιδεία, θα μορφωθούν οι γυναίκες περισσότερο. Έτσι θα προστατεύεται καλύτερα η γυναίκα στις χώρες αυτές. η συνεργασία και ανάπτυξη με τον ανθρωπιστικό παράγοντα πρέπει να είναι πράγματα τα οποία να υπάρχουν στις συμφωνίες που κάνουμε με τις εν λόγω χώρες που παραβιάζουν τα δικαιώματα των γυναικών. Και όχι μόνο. Πορνεία. Πώς να καταλήξουμε σε ευρωπαϊκή λύση. Εγώ συμφωνώ με τον κοινό στόχο Κοινοβούλιο και διάφορες χώρες μέλη, Συμβούλιο της Ευρώπης. Η κατάσταση όμως στις χώρες μέλη είναι πολύ διαφορετική από χώρα σε χώρα. Χρειάζονται διμερείς συνομιλίες. Αναφέρθηκα στην πορνεία σε σχέση με την βία σε βάρος των γυναικών. Το θέμα της πορνείας το βάζω πάντα με την βία σε βάρος των γυναικών. Υπάρχει ένα πρόγραμμα πολύ ενδιαφέρον. Θέλουμε να κάνουμε και κοινωνική δουλειά επιτόπου. Να βοηθήσουμε δηλαδή ψυχολογικά, υλικά. Η εκπαίδευση επίσης, συναισθηματική παιδεία είναι πολύ βασικό να παρέχεται από τις πρώτες τάξεις του σχολείου γιατί έτσι προωθείται η ιδέα της μη κυριαρχίας του ενός φίλου πάνω στο άλλο και βοηθάει να αντιληφθούν την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών από μικρή τα γόρια και τα κορίτσια. Σίγουρα θα έχω αφήσει πολλά απ' έξω, αλλά κοιτάω ότι πέρασε η ώρα, οπότε θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο. Μάλιστα αύξηση της απασχολήσεως των γυναικών. Ασφαλώς και είναι προτεραιότητα και πρέπει να είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες μιλούμε πολύ για την ε, απασχόληση των γυναικών, για την οικονομική τους ανεξαρτησία. Και μία από τις προτεραιότητες της λουξεμβουργικής κυβερνήσεως θα είναι και ο αγώνας κατά της φτώχειας παιδιών και γυναικών. Διότι με την αύξηση της γυναικείας απασχολησιμότητας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα αυτό. Τώρα, η οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών επίση επίσης πολύ σημαντική. Όπως είπα, αυτά τα δυο συμβαδίζουν. Η πρόσβαση δηλαδή στην αγορά εργασίας, πρόσβαση σε ε, αδιαμήτρότητας, επίσης αδιαπατρότητας για τους άντρες. Αυτά όλα θα βοηθήσουν για να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας η γυναίκα. Επίσης, κατάλληλη παιδική σταθμή και νηπιακή σταθμή κτλ. Όλα αυτά είναι σημαντικοί παράγοντε έτσι ώστε να μπορούν οι γυναίκε να βρουν δουλειά, να μπορέσουν να δουλέψουν επίση σε γαλήνη πνεύματο, χωρί να, να τρώνε οι έγνοιε του για το τι γίνεται το παιδί την ώρα που αυτέ εργάζονται. Όπω είπε η συνάδελφό μου Μούτ, η άδεια μητρότητα μα βρίσκει απόλυτα σύμφωνη, σα υποστηρίζουμε 20 εβδομάδε έχουμε εμεί άδεια μετρότητα στο Λουξεμβούργο και θεωρούμε ότι πράγματι θα πρέπει να υιοθετηθεί και από όλου. Είμαστε λοιπόν στο πλευρό σας για το διάβημα αυτό. Δεν αρκεί βέβαια να μιλούμε μόνο για άδεια μητρότητα. Πρέπει να μιλήσουμε και για άδεια πατρότητα και για γονική άδεια. Στο Λουξεμβούργο προχωρούμε τώρα σε αναδιατύπωση των αδειών αυτών, διότι για την ώρα οι άνδρε έχουν υπερβολικά μικρέ άδειε πατρότητα. Προσπαθούμε λοιπόν να τι κάνουμε πιο εύκαμπτε τι ρυθμίσει αυτέ και επομένω πιο, πιο αποδοτικές και πιο ενδιαφέρουσε για του άνδρε. Είμαι θα βέβαιε ότι πολύ περισσότεροι άνδρε θα επωφεληθούν από τι διατάξει αυτέ, κάτι το οποίο θα ωφελήσει και τι γυναίκε και του άνδρε στην πρόσβασή του στην αγορά εργασία. Η άδεια μητρότητα βέβαια είναι υπόθεση του Υπουργείου Εργασίας Είμαι βέβαια ότι στο Συμβούλιο Υπουργών θα τα πούμε τα πράγματα αυτά την Παρασκευή, θα τους μεταφέρουμε δηλαδή τόσο ακούσαμε σήμερα εδώ, διότι η Υπουργεία Εργασίας, η Υπουργεία Ισότητας και εγώ, Υπουργείο μάλλον Εργασίας Ισότητας και εγώ προσωπικά, θα συνεργαστούμε για να ανταλλάξουμε απόψεις, να προωθήσουμε τις άδειε που προανέφερα και σε άλλες χώρες. Σχετικά με τους Ρώμα. δεν αρκεί να οργανωθεί μια ετήσια επέτειος. Δεν αρκεί. Πρέπει και στα σχολικά προγράμματα των ε, παιδιών να μπουν, να μπει η ιστορία των Ρωμά, η οποία είναι αναπόσπαστο μέρος της δικής μας ιστορίας. Και τα νεαρά παιδιά του σήμερα είναι οι αυριανοί ενήλικοι. Αυτά πρέπει να μπουν στα σχολεία της Ευρώπης. Έχει πρωταρχική σημασία. Άκουσα επίσης σχετικά με γυναίκες από διάφορες ε, εθνικότητες. Επίσης είναι πολύ σημαντικό. Εμείς δεν ρωτούμε ποια είναι η θρησκεία σου, ποια είναι η εθνική σου καταγωγή, η εθνοτική σου καταγωγή. Πρέπει να μπορέσουμε να εντάξουμε, να ενσωματώσουμε όλες τις γυναίκες, όλες τις γυναίκες της κοινωνίας μας. Ανεξαρτήτως προελεύσεως. Να ενισχύσουμε δε και τις κοινωνίες εκείνες όπου δεν υπάρχει αυτή η νοοτροπία ισότητας να συμβάλλουμε ώστε να αντιμετωπίσουν οι κοινωνίες αυτές τις γυναίκες τους με ισοτιμότερο τρόπο με τους άνδρες. Πράγματα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε. Να ρίξω μια ματιά μου πως λησμόνισα τίποτα. Οι δράσεις κατά των διακρίσεων επίσης είναι σημαντικές. Είναι σημαντικό να εργαστούμε περισσότερο για την εξάλληψη των διακρίσεων και βεβαίως και υπέρ της πολυφωνίας, της ποικιλία τις ποικιλομορφία, να δούμε τα προβλήματα, αλλά όχι μόνο ως προβλήματα, να τα δούμε και ως ευκαιρίες. Έχουμε διαφορετικές εθνικές καταγωγές, διαφορετικές θρησκείες και ούτω Αυτά μπορούν να είναι και ισχυρά σημεία, όχι μόνο αδυναμίες. Να συζητήσουμε τα θέματα αυτά, να δούμε πώς μπορούμε να ζητήσουμε και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας βοηθήσει ώστε να καταστούν γνωστά τα προβλήματα αυτά. Διότι ο φόβος απέναντι στον άλλο τελικά προέρχεται από το ότι δεν τον γνωρίζουμε. Αν τον γνωρίσουμε καλύτερα θα μειωθεί ο φόβος. Να μάθουμε, να διδάξουμε στους πολίτες μας να γνωρίσουν καλύτερα τον άλλο και να αποδεχτούν την διαφορά. Είτε αυτή είναι διαφορά θρησκευτικών πεπιθήσεων, είτε γενετήσιου προσανατολισμού η οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επαναλαμβάνω ότι η Επιτροπή μας θεωρεί ότι είναι ανάγκη να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Λουξεμβουριανή Προεδρία. Πρώτα απ' όλα το βλέπουμε όταν κάποιος αναλαμβάνει μια δέσμευση και όταν δείχνει ευαισθησία στα θέματα της ισότητας των δύο φύλων. Οπότε σας εύχομαι κάθε επιτυχία αυτούς τους μήνες, γιατί δικές σας επιτυχίες θα είναι και δικές μας. Ολοκληρώνουμε εδώ τις εργασίες της Επιτροπής μας και πάλι ευχαριστώ τους δύο υπουργούς που συμμετείχαν στην ανταλλαγή αυτή απόψε. Ευχαριστώ. Les recuerdo que ahora continuamos en la reunión de coordinadores posteriormente. Συνεχίζουμε με τη συνεδρία των συντονιστών.